Please take a seat. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε καθίστε και καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας, να αρχίσουμε τις συνομιλίες μας. Έχετε την ημερήσια διάταξη, τροποποιήσεις δεν έχουν προταθεί, εγκρίνεται. Σας παραπέμπω στο Cont News, έχουμε web streaming, ε, Πρόεδρε, για την ημερήσια διάταξη υπάρχουν δύο σημεία στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Το ένα, να καταγραφεί στα πρακτικά η διαμαρτυρία μας, το ότι γίνεται ψηφοφορία μία Δευτέρα στις 3 το απόγευμα που επανειλημμένα έχουμε πει ότι είναι πολύ κακή μέρα γιατί πολλοί βουλευτέ έρχονται από μακρινέ χώρε και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν ακριβώ εδώ στι 3 γιατί δεν έχουν καλή ανταπόκριση και πόσο μάλλον μετά το Στρασβούργο. Και δεύτερο, να σας ρωτήσω το εξή. Βλέπω ότι στο σημείο 8 έχουμε την παρουσίαση της συγγήτριας, ε, της κυρίας ε, Χολμάιερ, ε, και ήθελα να ρωτήσω, είναι της Επιτροπής Budget, ε, γιατί λοιπόν παρουσιάζει την ε, γνωμοδότησή της εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί μας παρουσιάζει η συγγήτρια αυτή την γνωμοδότηση και παρουσιάζει αυτή την γνωμοδότηση εδώ αντί να την παρουσιάσει δική της Επιτροπή. Δεν είναι λοιπόν δική μας εισηγήτρια, αλλά προέρχεται από την Επιτροπή Υπερπολογισμών. Για τις ψηφοφορίες. Θεωρήσαμε ότι όποια δυσκολία είναι ίδια για όλες τις ομάδες και άρα έχουμε ισότητα δυσκολιών ούτως υπήρει. Πάντα κοιτάμε να κάνουμε ψηφοφορίες το απόγευμα για να έχουμε το χρόνο να Ολοκληρώνουμε την ημερήσια διάταξη και δεδομένου ότι έχουμε και τις απαλλαγές και τα περιφερειακά θέματα δεν είναι βέβαιο ότι θα προλαβαίνουμε. Προσπαθούμε λοιπόν πάντα να δίνουμε την ευκαιρία στους συναδέλφους να είναι παρόντες. Για το 8 η Επιτροπή των Προϋπολογισμών έχει ψηφίσει αυτή την έκθεση, μόλις μάλιστα, Υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και γι' αυτό η κυρία Χολμάιερ στην συνεδρία της Επιτροπής των Προϋπολογισμών ζήτησε να το παρουσιάσει, να το εκθέσει στη δική μας Επιτροπή και γι' αυτό το περιλάβαμε στην ημερήσια διάταξη. Είναι θέμα ελέγχου του προϋπολογισμού και πρέπει να μας απασχολήσει οπωσδήποτε και αμέσως. Γι' αυτό το περιλάβαμε στην ημερήσια διάταξη και φαντάζομαι ότι μπορείτε και δείξετε κατανόηση στην παρουσίαση του θέματος από την κυρία Χολμάιερ. Θα αντιληφθείτε περί τίνος πρόκειται. Σημείο 3. Ψηφοφορία. Γνωμοδότηση του κυρίου Σαββάρμα. Πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλει η έκθεση της Επιτροπής των Προπολισμών. Θέλει ο κύριος Σαββάρμα να πει κάτι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με ικανοποίηση σημειώνω ότι είναι αρκετοί οι συνάδελφοι που είναι εδώ παρόντε, έστω και δεύτερο απόγευμα. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και την παρουσία μας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση. Ας ψηφίσουμε μία μόνο τεχνικού τύπου διόρθωση στον κατάλογο ότι αν εγκριθεί η τροπολογία περιθμών 6 θα καταπέσει η 9. Εάν εγκριθεί η 6 καταπίπτει η 9. Και για το ΕΛΚ υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές στο κατάλογο ψηφοφοριών, αλλά δεν θα σας κουράσω με αυτά. Καλώς λέει η Πρόεδρος, ψηφίζουμε. Έχει δυναμηθεί ο κατάλογος. Τροπολογία θυμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη καλά ας επαληθεύσουμε την 4 Επαληθεύσαμε λοιπόν και απερίφθη 8 ψήφι υπέρ, 8 κατά. Υπαριθμόν 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 6 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 6 παρακαλώ. Πέρασε. Απερίφθη. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε την 8. Όχι, εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος, συγγνώμη. Εγκρίνεται. Πέρας της επαλήθευσης. 9. Και είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε το 15 πέρας εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 17 χωρί ψηφοφορία, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε την 28 πέρας απερίφθη 29 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 50 διαγραφή ε, έως 53 υπέρ κατά 50 έως και 53 σε μια ψηφοφορία επαληθεύουμε πέρας της επαλήθευσης εγκρίνονται 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη επαληθεύουμε 54 πέρας απερίφθη 55 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56 και 57 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε 56-57. Ναι, είναι το ίδιο, η ίδια ψηφοφορία με την 55. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας, απερίφθη. 58 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 59 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη επαληθεύουμε την 59 πέρας απερίφθη 60 χωρίς φορεία τεχνική διόρθωση 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές 66 παρακαλώ επαλήθευση όλο και έρχονται οι συνάδελφοι πέρασε της εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68-69 μαζί σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 70 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 70 επαληθεύουμε πέρας απερίφθη 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 73 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 74-75 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 76 κατά αποχές απερίφθη 77 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απερίφθη η 80 σε δύο τμήματα με προφορική τροπολογία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε πρώτο τμήμα της 80 νομίζω ότι έχει απορριφθεί Πέρας. Εγκρίνεται. Καλά κάναμε και επαληθεύσαμε. Προφορική τροπολογία. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Επαληθεύουμε λοιπόν 80 δεύτερο τμήμα. Επαληθεύουμε δεύτερο τμήμα της 80. Και εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Να επαληθεύσουμε. 84. με διαγραφή. Πέρας απερίφθη. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 87 σε δύο τμήματα υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε το δεύτερο της 87. πέρας απερίφθη 88 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 90 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε είναι 90 90 πέρας απερίφθη 91 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 92 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 94 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 95 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη μαζί με την 96 και 97 μαζί υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 98 να επαληθεύσουμε λοιπόν την 97. Ναι, δεν ήταν σαφής ο κατάλογος των ψηφοφοριών. Πέρασε ψηφοφορία, σε 99 υπέρ. Όχι. 98 τώρα. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 103 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 104 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 105 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 106 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 109 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη. Να επαληθεύσουμε την 109. 109. Πέρας. Απερίφθη. Γνωμοδότης το σύνολό της. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 10 ψήφι υπέρ και 8 κατά. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στεχόφσκι είναι ο εισηγητής. Θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια παρατήρηση.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 Πέρα ψηφοφορία, απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Καταπίπτει. 19. Επίση καταπίπτει. 20. Επίσης 21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22. 23 και 24. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε βεβαίως. Ψηφίζουμε την τροπολογία 26. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 έχει, την έχουμε διεκπαιρεώσει με τη συμβαστική 2. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ναι, να το έλεγξουμε. Επαληθεύουμε την τροπολογία 33. Πέρας της εφορίας. Απορρίπτεται σαφώς. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 διεκπαιρεώθηκε. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. 41 νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά για να είμαστε σίγουροι. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 44 καλύπτεται από την συμβαστική 1. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική να την ελέγξουμε. Μάλιστα, ελέγχουμε την 3. Συμβαστική πρόταση 3. Επαληθεύουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέλος ψηφοφορίας λοιπόν. Και ψηφίζουμε την ε, πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Τελική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 17 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έτσι. Alles klar, danke. Bei Tagesordnungspunkt Nummer 4. Φτάνουμε στο σημείο 5 της ημερής της διάλεξης. Ακρόαση της Επιτρόπου Κρέτου. Πέντε λεπτά νωρίτερα τελειώσαμε, αλλά νομίζω ότι η Επίτροπος ήδη έχει έρθει. Να δει κάποιος Πότε να υπολογίζουμε παρακαλώ ότι θα έρθει η κυρία Επίτροπος, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχωρούμε λοιπόν. Να καλωσορίσω την Επίτροπο αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική. Και βεβαίως να καλωσορίσουμε και την κυρία Ιβάνοβα, το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγχαρητήρια για, ε, ε, για τον επαναδιορισμό σας στην ε, θέση σας από την προηγούμενη συνεδρίαση του στο Στρασβούργο. θα πάρετε εσείς πρώτο λόγο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κύριε συγητά, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα και τις συστάσεις για το κεφάλαιο 6 της ετήσιας εκθεσής μας για το έτος 2016. Το κεφάλαιο αυτό σχετίζεται με τον τίτλο 1B του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και καλύπτει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Επίσης, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική και ε, σχέση που είχαμε, πολύ επικοδομητική καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία, και ξεκινώ κατευθείαν με τα βασικά δεδομένα για του ελέγχου που έχουμε κάνει για παρατυπίε. Για το 2016 ο πληθυσμό που ελέγχθηκε ήταν 36 ε, δισεκατομμύρια. Από αυτό 21 δισεκατομμύρια σχετίζονται με το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξη και άλλα 17,5 με το Ταμείο Συνοχή και 8,1 δισεκατομμύρια με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η διαχείριση των τομείων αυτών είναι κοινή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και το 2016 ήταν το τελευταίο έτο κατά το οποίο όλε οι πληρωμέ ε, ελέγχθηκαν που σχετίζονται με, το 2010, ε, με την προγραμματική περίοδο 2013-2017. Για από του ελέγχου μα, ελέγξαμε ένα αντιπροσωπευτικό ε, δείγμα 180 συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων 12 ε, δημοσιονομικών εργαλείων τη κοινή αυτή διαχείριση. Το ε, επίπεδο λάθο ήταν 4,8%. Είναι χαμηλότερο από το 5,2 βεβαίως ε, που είχαμε το προηγούμενο έτος, αλλά παραμένει ιδιαίτερος υψηλό και σίγουρα πάνω από το, ε, από το επίπεδο που θα θέλαμε που είναι 2%. η βάση για το, για το βαθμό λάθους είναι τα 25 λάθη που ποσοτικοποιήθηκαν από το δείγμα μας. Τα ε, βασικά είδη λαθών τον, του τίτλου αυτού σε, με βαθμό σημασία είναι τα μη επιλέξιμα ποσά ε, σε σχέση με τι δηλώσει κόστου 42%, σοβαρά λάθη στι δημόσιε προμήθειε 30% και μη επιλέξιμες δραστηριότητες και project 28%. Θα ήθελα επίσης να σα επιστήσω την προσοχή, κύριε Πρόεδρε, σε διάφορα σημαντικά στοιχεία, τα οποία επίσης τονίζουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Να ξεκινήσω με τι απλουστεύσεις. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε εξετάσει 135 συναλλαγές που χρησιμοποίησαν απλοποιημένες ε, επιλογές για την ε, δήλωση δαπανών, 10% ε, δηλαδή των συνολικών συναλλαγών. Και βρήκαμε μηδέν ε, προσωπικοποιήσιμα λάθη σε αυτές τις 135 συναλλαγές που δείχνει ότι τα project που χρησιμοποιούν απλουστευμένους τρόπους ε, δήλωση δαπανών ε, κάνουν λιγότερα λάθη σε σχέση με αυτούς που έχουν επιστρεφόμενα έξοδα. Για, το, για την προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020 τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να κάνουν ευρύτερη χρήση αυτών των επιλογών των απλουστευμένων για το τομέα της συνοχής. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο του κεφαλαίου αυτού είναι η επέκταση της ε, περίοδου επιλεξιμότητας για, την, για τα δημοσιονομικά εργαλεία. Έχετε, το έχετε συζητήσει και εσείς, το έχουμε συζητήσει και εμείς πολλές φορές. Συνοπτικά, αυτό που μπορώ να σας πω είναι τον Απρίλιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει την περίοδο αυτή για τα δημοσιονομικά εργαλεία από, 30, από την 31η 31 η δεκεμβριου 2015 στο 31η Δεκεμβρίου 2017 αντί να κάνει πρόταση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να τροποποιήσει τον σχετικό κανονισμό. Είναι ο τρίτος χρόνος αυτός ε, στη σειρά που τονίζουμε ε, εμείς ως Ελληνικό Συνέδριο αυτή την ε, πτυχή της νομικής ερμηνείας και υπολογίζουμε ότι η αξία των αγγίσεων και των πληρωμών που γίνονται σε αυτή τη διαβριμένη περίοδο φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρ' αυτά δεν έχει συμπεριληφθεί στο βαθμό λάθους γιατί είναι άπαξ ευρήμα, το οποίο δεν επηρεάζει καθόλου τον ευρωπαϊκό προεπλογισμό στο σύνολό του και δεν επιτρέπει συγκρισιμότητα με προηγούμενα έτη. Άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι ο καθορισμός των, των ε, κρατικών αρχών που είναι υπεύθυνα για τα ε, κονδύλια αυτά. Για πέμπτο έτος ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, καθυστερήσεις από την, ε, στα πλαίσια αυτής της προγραμματικής περίοδου μέχρι το 2020. Μέχρι το Μάρτιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τους τελικούς λογαριασμούς με δαπάνες που καλύπτουν το 0,7% του προϋπολογισμού που είχε οριστεί για όλη την προγραμματική περίοδο. Μέχρι τα μέσα του 2017 οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προπολογισμού ήταν μεγάλες και ήταν το ίδιο με την ε, περίοδο 2013-2017. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι τα κράτη-μέλη είχαν ορίσει μόνο 77% των αρχών που είναι υπεύθυνε για την πολιτική συνοχή και τη διαχείριση των κονδυλίων μέχρι το τέλος του 2016. Άλλο ένα σημαντικό σημείο του ελέγχου μας είναι η εξέταση των ε, ε, εργαλείων της Κομισιόν για, το για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το νομικό πλαίσιο αυτής της περίοδου εισάγει έναν αριθμό βελτιώσεων, όπως οι ε, απαλλαγές αιτήσει, το κλείσιμο των λογαριασμών, τα πακέτα ασφάλισης και μια συστηματική διατήρηση του 10% κάθε ενδιάμεση πληρωμή, καθώ επίση και ε, καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων. Η βασική προπόθεση για την εξαίρεση από του λογαριασμού και για την ε, δημοσίευση των αιτήσεων λογαριασμών είναι ότι το εναπομείναν ποσό από τα κράτη-μέλη και τι αρχέ του που λαμβάνουν υπόψη βεβαίως όλες τις δημοσιονομικές διορθώσεις, παραμένει κάτω από το 2%. Εμείς ως ελεκτικό συνέδριο λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις αλλαγές για το, στο σχεδιασμό των, των, των ελέγχων μας για το 2017 και ως πολιτικό εγχείρημα θα κάνουμε ε, μια δοκιμή στην, ε, στον τομέα της συνοχής έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερη χρήση των ε, πληροφοριών που μας δίνουν οι ελεκτικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να παράσχουμε στεγανά και αξιόπιστα ε, αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια των ε, δραστηριοτήτων μας. Ε, είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά κονδύλια να δαπανώνται με βάση τους κανόνες. Είναι πρώτη προϋπόθεση αυτή για να έχουμε αποτελέσματα. Το δεύτερο όμως σημαντικό βήμα είναι να επιτύχουμε την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια και βεβαίως εξοικονόμηση πόρων. Ε, για τρίτη χρονιά φέτος ε, έχουμε ένα ξεχωριστό κομμάτι στο κεφάλαιο αυτό που έχει να κάνει με την αξιολόγηση της ε, αξιοπιστίας του, του δείγματός μας. Ξέρουμε ότι ο σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης απόδοσης είναι πιο σημαντικός για την περίοδο 2014-2020. Ας πούμε, οι ελεκτικές αρχές στα κράτη-μέλη τώρα πρέπει να εξετάζουν την ευθύνη των δεδομένων και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να επιβληθούν ε, ποινέ σε περίπτωση που υπάρχουν ε, ίσως ε, σημασίες αποτελέσματα από τα κράτη-μέλη. Για το 2020-30 είναι σημαντικό να, να σημειώσουμε ότι το νομικό πλαίσιο δεν υποχρεώνει τις προγραμματικές αρχές να ορίσουν δείκτες ε, ανά project. Γι' αυτό είδαμε ότι μόνο ένα τρίτο των 168 project που εξετάστηκαν είχαν ε, και σύστημα αξιολόγησης απόδοσης συνδέοντας δηλαδή το αποτέλεσμα με τους στόχους που είχε θέσει το πρόγραμμα. Επιπλέον, έχουμε καταγράψει κάποιες αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη έχουν σχεδιάσει τα συστήματα αυτά και σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο project. Παρά αυτά τα λάθη στην διαχείριση των project είναι σημαντικό να πούμε ότι σχεδόν όλα ε, δηλαδή 92% των project που ελέγχθηκαν ε, πέτυχαν τους στόχους που είχαν θέσει είτε ολικός είτε μερικός. Επίσης, Κάνουμε τρεις συστάσεις σχετικά με το, με το κλείσιμο του ε, επιχειριστικού προγράμματος ε, μέχρι το 2017 και για τους υπολογισμούς του εναπομείναντος ε, βαθμού λάθους για την περίοδο 2014-2020 και για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να ενισχυθεί η ε, επικέντρωσή μας στην απόδοση, κυρίως δηλαδή δέσμευση των πληρωμών με την απόδοση και όχι απλώς αποζημίωση δαπανών. Όλες αυτές οι συστάσεις έχουν γίνει ε, αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήγοντας να πω ότι η πολιτική συνοχή παραμένει μία από τι βασικέ πολιτικέ επένδυσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πολιτική όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει την προστιθέμενη αξίματα, δείχνοντα αποτελέσματα που είναι ορατά από όλου του Ευρωπαίου πολίτε, εάν εφαρμοστούν τα προγράμματα σωστά. Ελπίζω τα συμπεράσματά μα και οι συστάσει μα να έχουν αξία και για εσά και να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, κυρίως για τη δουλειά της Επιτροπής σας, αλλά και για τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Εισηγητά, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το κεφάλαιο και καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε για τα περιφερειακά. 78 ερωτήσεις έχουμε υποβάλει. Ευχαριστούμε και εσά και την ομάδα σα για τι απαντήσει που μα δώσατε και έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you, ναι, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Σεγητά, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ε, κυρία Ντίνα από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, κυρίε και κύριοι. Καταρχήν, ε, θέλω να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για τα θετικά νέα ε, φέτος για την ε, ειδική γνωμοδότηση για τις πληρωμές του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική συνοχές. Ε, μειώθηκε το ποσοστό λάθους για πέμπτο έτος κατά σειρά και τώρα είναι κάτω του 5%. Με άλλα λόγια, πάνω από 90% των πληρωμών, 95% των πληρωμών ήταν χωρίς λάθος. Αυτό μας δείχνει τη βελτίωση της διαχείρισής μας ε, και των συστημάτων ελέγχου και του συλλογικού έργου στο να μειώνεται το ποσοστό λάθους ε, με το πέρασμα του χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και ιδίω την Επιτροπή ΚΟΝΤ που μας δίνει την υποστήριξη για την επίτευξη όλων αυτών. Τώρα είμαστε κοντά στο κλείσιμο της διαδικασίας ε, των προγραμμάτων 2007-2013 που καλύπτονται από αυτή την ετήσια έκθεση θα κλείσει το πρόγραμμα μόνο αν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν παραμένουν λάθη. Ε, η Κομισιόν έχει χρησιμοποιήσει προληπτικά μέτρα και έχει κάνει χρηματοοικονομικές διορθώσεις ε, στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε διασφαλίζοντας ότι το λάθος παραμένει κάτω το 2%. Αυτό θέλουμε να ισχύει και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Φυσικά μεγαλύτερη λογοδοσία θα έχουμε από τις αρμόδιες αρχές και θα ε, παρακρατούμε το 10% των ε, πληρωμών ε, μέχρι τον πλήρη έλεγχο και φυσικά μέχρι να γίνουν και οι απαραίτητες οικονομικές διορθώσεις πρώτο ποσοστό λάθους που αναφέρθηκε από τα κράτη-μέλη είναι πολύ κάτω του 2%. Κυρίες και κύριοι, ε, μπορώ να κατανοήσω εδώ τις ανησυχίες ε, του Προεδρού, του κυρίου Λένε, ότι οι άνθρωποι θέλουν και έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ε, ποια είναι η αξία των χρημάτων τους. Φυσικά η συμμόρφωση με τους κανόνες, όπως είπε και η κυρία Ντίνς, ε, είναι μόνο ε, το ίμιση του παιχνιδιού. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, και μεγάλες προσδοκίες από την Επιτροπή Κοντ να δείξει ότι χρησιμοποιούνται πολύ σωστά τα χρήματα του φορολογουμένου και ότι έχουμε επιδόσεις, έχουμε τις εκθέσεις εφαρμογών για κάθε πρόγραμμα και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε υπερβεί και τους στόχους. Τώρα θέλω να αναφερθώ και στην έκθεση πολιτικής του 7ου προγράμματος. Βλέπουμε να μειώνονται πάλι τα χάσματα μετά από μια περίοδο που ακολούθησε τη χρήση έχουμε ανάκαμψη των, ε, της απασχόλησης, των θέσεων εργασίας, αν και χρειάζονται επενδύσεις ε, στην καινοτομία, στις υποδομές ε, και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική συνοχής έχει βοηθήσει πολύ για να ξεπεράσουμε την ύφεση ήταν ε, η κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης τα τελευταία τρία χρόνια. Είχαμε χρηματοδότηση κατά 85% μέσο όρο σε δημόσιες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό το ποσοστό φτάνει σε πάνω από 40% ε, για κράτη-μέλη όπως η Κροατία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Λιθουανία. Έτσι λοιπόν ο αντίκτυπος ε, της ε, πολιτικής συνοχής στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι σημαντικός και τα αποτελέσματα των επενδύσεων είναι μακροπρόθεσμα. Για το σημερινή χρηματοοικονομική περίοδο έχουμε υποστηρίξει 1,1 εκατομμύρια μικρές και μεσές επιχειρήσεις, 60 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύονται στην ψηφιακή οικονομία. Ε, φτάνουμε περίπου σε 50 εκατομμύρια νοικοκυριά που έχουν ευρυζωνικό διαδίκτυο. Επίσης επενδύουμε στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση του κοινωνικού επικλεισμού, στη βελτίωση ε, των δημόσιων μεταφορών ε, μέσω της βελτίωσης του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Τα ωφέλη των προγραμμάτων μας ε, υπερβαίνουν την οικονομική και κοινωνική διάσταση. Η πολιτική συνοχή βελτιώνει και τη διακυβέρνηση στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Ε, βλέπουμε ε, μια βελτίωση των ε, επενδύσεών μας. Ξέρετε ότι με την εξάντε μέσω της φιούς εξειδίκευσης, με την εστίαση στις επιδόσεις, πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι ισχύει η αιρεσιμότητα εξάντη για όλα τα προγράμματα με κάποιες εξαιρέσεις όπου εφαρμόζουμε τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό. Δηλαδή ότι μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις δεν προβαίνουμε στις πληρωμές. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα και τις επενδύσεις κάθε χρόνο ε, έχουμε δημοσίευση ε, των σχετικών δεδομένων μέσω της πλατφόρμας. Ε, μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα της ΓΔΡ βλέπουμε τους στόχους για κάθε πρόγραμμα, περιφέρεια και κράτος μέλος. Ξέρω ότι κυρίως ε, αυτή η Επιτροπή ανησυχεί για το επίπεδο των πληρωμών μέχρι τώρα για την περίοδο 2014-2020. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων σημειώνει καλή πρόοδο επιτόπου. Είμαστε στο 44% για την πολιτική συνοχής ε, και ε, για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο ως προς την απορρόφηση. Όμως συμφωνώ μαζί σας ε, ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο επίπεδο των πληρωμών και Πιστεύω έχουμε αρκετούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην κατάσταση. Καταρχήν η καθυστερημένη υιοθέτηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου καθυστέρησε όλα τα προγράμματα και ο κανόνας νη ε, συν τρία έχει μειώσει την πίεση για την καταβολή των πληρωμών ε, και πρέπει να δούμε αν ε, θα επανέρθουμε στον νη συν 2 γιατί, παραδείγματο χάρη από φέτο, ε, είναι πολύ σημαντική πίεση για τα κράτη-μέλη. Και πιστεύω ότι ο φόβος ε, των κρατών μελών ε, για τις καθαρές χρηματοοικονομικές διορθώσεις στους ετήσιους λογαριασμούς έχει παίξει ρόλο στις καθυστερήσεις. Πάντως, θέλω να σας καθησυχάσω για το εξής ο διορισμός των αρχών ε, για να στέλνουν ε, ε, στην Κομισιόν τις απαιτήσει δεν είναι πλέον θέμα. Έχουμε τώρα διορίσει το 90% των αρχών για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τα τέλη του έτους και για την πολιτική συνοχή πρέπει να, πάμε περαιτέρω, να προχωρήσουμε περαιτέρω στην απλούστευση, καθώς η ομάδα υψηλού επίπεδου, ε, οι συστάσεις αυτής της ομάδας και ο κανονισμός Omnibus είναι πολύ σημαντικά εργαλεία και εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είστε τώρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία ως συνομοθέτες και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. για μετά το 2020 είμαι υπέρ μεγαλύτερης απλούστευσης, πιο ριζοσπαστικής απλούστευσης, είναι απαραίτητη. Πρέπει να δούμε κάθε πτυχή της πολιτικής και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να απλουστεύσουμε πάρα πολύ, ενώ θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της πολιτικής που λειτουργούν καλά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να βρούμε την ορθή ισορροπία μεταξύ της συνέχειας και της μεταρρύθμισης. Θα παρουσιάσουμε τις νομοθετικές προτάσεις ε, για την πολιτική συνοχή μετά το 2020, μετά την ε, υποβολή του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου τον επόμενο Μάιο. Αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι είναι ικανή να απαντήσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η πολιτική συνοχής ε, έχει πολύ σημαντική συνεισφορά. Είναι μοναδική γιατί συνδυάζει την ευρωπαϊκή και εθνική προοπτική με την περιφερειακή και τοπική προοπτική. Επίσης, αυτό είναι το μέλλον για την εξειδίκευση για να μπορέσει να μεγενθηθεί η κάθε περιφέρεια και η πολιτική συνοχή πρέπει να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική για όλες τις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, το πιστεύω μόνο εγώ αυτό ε, και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αυτής της εβδομάδας αλλά και όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν με την άποψη αυτή. Και φυσικά βασίζομαι στην συνεχή υποστήριξή σας για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των ε, σημερινών προγραμμάτων και να κάνουμε πιο αποτελεσματική την πολιτική στο μέλλον. Έχω, ξέρω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία καθ' όλα αυτά τα έτη. Ευχαριστώ. Έχουμε όντω κάποιε ερωτήσει. Φαντάζομαι. Ο εισηγητή ήταν ο πρώτο. ο κύριο Τσέλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς την κυρία Ιβάνοβα. και την ομάδα των συνεργατών του Λεκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση της έκθεσης ε, του Λεκτικού Συνεδρίου για το 1Β του προπολογισμού στη διαδικασία απαλλαγής για το 2016 και τις σχετικές επαληθεύσεις. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο Κρέτσου και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακών, Περιφερειακής Πολιτικής για τις απαντήσεις στις 76 ερωτήσεις. Θα συμφωνήσω και με την κυρία Ιβάνοβα και με την κυρία Κρέτσου. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Διαρθρωτικά Ταμεία είναι το κατάλληλο μέσον και για την υποστήριξη των επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση στη διάθεση των κρατών μελών των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός αλλά αφετέρου ταυτόχρονα πρέπει και να καθιστούν ορατή, την, ε, ορατό το μέλημα για συνοχή Θέλουμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία και όπου υπάρχουν ανησυχίες, αδυναμίες στις οικονομικές εξελίξεις. Θέλουμε από κοινού και με βάση βέβαια και την αρχή της αλληλεγγύης να τις αντιμετωπίσουμε. Εδώ λοιπόν επισημαίνω έχοντας μια προϋπηρεσία περίπου δύο ετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι όταν ε, γίνεται λόγος για απασχόληση και ανάπτυξη μετά την ε, έναρξη της κρίσης του 2008 θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες ε, στις, στη συνοχή και να ενισχύσουμε τα διευθυντικά ταμεία. Τώρα όμως αυτή η φωνή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο από την κυρία Κρέτσο και από τον Επιτροπό για τον Προπολογισμό Αρμόδιο, τον κύριο Έτιγκερ, φαίνεται να είναι πιο ε, χαμηλόφωνη. Ναι, μεν μένει το Διευθυντικό Ταμείο, αλλά ταυτόχρονα ακούγονται άλλες φωνές που λένε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν άλλα μέσα συμπληρωματικά, όπως Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΤΣΕ. Και όντως μπορεί καταρχάς να είναι πηγή αισιοδοξία στο γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος κατά την εκτέλεση της περιφερειακής πολιτικής και του Ερωτικού Ταμείου έχει πέσει να είναι στο 4,8% αλλά δεν πρέπει και να ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε επιμερισμένη διαχείριση. Επιτροπή, κράτη-μέλη, σε ένα βαθμό μάλιστα και αρχές αρμόδιας διαχείρισης από τις περιφέρειες εμπλέκονται στη διαχείριση των ε, κονδυλίων αυτών ή και από άλλους τομείς μάλιστα. Πράγμα το οποίο έχει μάλλον περιπλέξει τις διαδικασίες. Άρα είναι ευπρόζεκτη κάθε μείωση του ποσοστού σφάλματος εδώ. Για το 2016 συγκεκριμένα, που, όπου σε απασχολεί η απαλλαγή, ε, πρόκειται για το τρίτο έτος της πολιετούς δημοσιονομικής περίοδου 2014-2020 επισημένο και από τη δική μου εμπειρία αλλά και από τα όσα έχω ακούσει και από αντιπροσωπείες από κρατημέλη στο τομέα της συνοχής ιδιαίτερος, όχι μόνο αλλά και από τις, προηγούμενες, από τις πρώην περιοχές στόχου 2 βλέπουμε ότι το 2016 έχουμε ακόμα κάποια ζητήματα σε σχέση με την ε, ολοκλήρωση, περαιτέρω επεξεργασία, εκτέλεση προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, 2006-2013 δηλαδή, και σχέδια ή προγράμματα της νέας ε, περίοδου ανάπτυξης, μπορεί ακόμη να μην έχουν καν ξεκινήσει. Και νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί στην επισήμανση για καθυστερήσει και ε, υπολοιπόμενη εκτέλεση ή υλοποίηση που αναφέρει και η κυρία Κρέτσου για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Σε αυτό πρέπει να γίνει βέβαια, πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Σε τι οφείλεται. Το αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο ότι στα τέλη του 2016 δεν ήταν ε, ακόμη, δεν είχαν διοριστεί όλες οι αρμόδιες για τη διαχείριση αρχές εγώ προσωπικώς διαπίστωσα ότι και πεπειραμένες υπηρεσίες διαχείρισης ή φορείς διαχείρισης πεπειραμένοι που είχαν και στο παρελθόν αναλάβει τέτοια έργα, ε, είχαν δυσκολία και ως προς τους διορισμούς, γιατί υπήρχαν ε, με τον νέο κανονισμό πλέον ε, να εκτελέσουν προϋποθέσεις και περαιτέρω διαδικασίες που είχαν συμπληρώσει και τα κράτη-μέλη στο διατακτικό, για να το πω ευγενικά. Και έτσι οι αρχές, οι οποίες ήταν αρμόδιες για την ε, διαδικασία του διορισμού και την επαλήθευση των ε, διαχειριστικών αρχών ή φορέων, τώρα έπρεπε και να επαληθεύουν με βάση αυτές τις νέες διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης. Έτσι λοιπόν και πεπειραμένες αρχές διαχείρισης ε, διαμαρτύρονται και μας λένε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου ε, δεν έχουν αποτέλεσμα ικανοποιητικό από τους, τις προσπάθειές τους. Και έτσι η εκτέλεση έργων και προγραμμάτων στη νέα αυτή προγραμματική περίοδο παρουσιάζει καθυστέρηση και αντίστοιχα μειωμένη, ε, μειωμένα ποσοστά απορρόφησης για την τρέχουσα προγραμματική ε, περίοδο, επαναλαμβάνω, σε προγράμματα ή έργα τα οποία έχουν να κάνουν με στρατηγικό σχεδιασμό. Πρόκειται για έργα τα οποία θα έπρεπε κανονικά να τα οποία ε, το 2016 ή δεν είχαν επαρκώς αναπτυχθεί ή έχουν καθυστερήσει. Και είπε και η κυρία Κρέτσου ότι για το 2017 περιμένει καλύτερες επιδόσεις, καλύτερη απόδοση και για την προγραμματική περίοδο του 2017 με τους νέους στόχους και τη στρατηγική 2020 και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχει παρουσιαστεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτό το σημείο. Εδώ πλησιάζει με δρασκελιές μεγάλες στο τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Θα δούμε αν θα μπορούσαμε στο τέλος του 2020 να έχουμε τη διαδικασία νήσιν που θα διευκολύνει τα κράτη-μέλη ως προς την αντιμετώπιση της ε, σύμπτωσης της ε, διοικητικής των διαφόρων προγραμματικών περιόδων ή αν θα πρέπει να περάσουμε σε άλλη διαδικασία για να επιταχύνουμε την ε, άντληση των ε, κονδυλίων στην ώρα τους. Είναι μια δουλειά την οποία θα πρέπει να κάνουμε εγκαίρως, μια συζήτηση πρέπει να κάνουμε εγκαίρως, γενικότερα στο πλαίσιο και τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής για τη δημοσίευση των ειδικών ε, συστάσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως θα μπορούσε να τη συμπεριλάβει από την επόμενη χρονιά στην τακτική της έκθεση. Έχουμε άλλωστε έγγραφα και απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρέχουσα έκθεση με το 7ο πρόγραμμα και την έκθεση για το 7ο πρόγραμμα που μπορεί να μας είναι χρήσιμες οι απαντήσεις αυτές και στη διαδικασία ε, απαλλαγής για το 2016 για τις, ε, για τις πιστώσεις οι οποίες ε, μπορεί να είναι σε κίνδυνο. Είναι το 2015-2016 λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω αν ο υπολογισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε υπολογισμούς με τα ίδια ποσά, εάν πρώτα βγάλουμε από το λογαριασμό μας κάποια ποσά τα οποία θεωρήσουμε ότι μπορεί να έχουν κάποιο σφάλμα, αλλά μετά ταυτόχρονα τα υπολογίζουμε ως καθαρά ποσά. δεν θα ήταν καλύτερο να μια διαφορετική και πιο απλή λύση. Επίσης, ε, από, τις, ε, από τους φορείς διαχείρισης των πιστώσεων ε, μαθαίνω ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες, έχουν πολλαπλασιαστεί οι διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου και έχουν και καταστεί πολύ πιο περίπλοκες. Έτσι λοιπόν και οι υπηρεσίε τη Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει πιστεύω να καταλήξουν σε ένα single audit concept ή principle. Θα πρέπει δηλαδή να επεξεργαστούμε μια ενιαία αρχή δημοσιονομικού ελέγχου έτσι ώστε η εκτέλεση των ερθωτικών ταμείων που πιστεύω εγώ τουλάχιστον και ελπίζω ε, ότι θα πρέπει στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής ε, μετά το 2020 και για την προσεχή προγραμματική περίοδο να είναι ακόμη στη διαθέση των κρατών μελών και των περιφερειών. Θα πρέπει λοιπόν έτσι να απλουστευτεί η διαχείρισή τους για τις αρχές εκτέλεσης. Αντί να έχουν τρεις διαφορετικούς δημοσιονομικούς ελεγκτές απέναντί τους Πράγμα που σε τελευταία ανάλυση με όλου του ελέγχου δεν του επιτρέπει να κάνουν τη δουλειά του στην ουσιαστική, δηλαδή την εκτέλεση των προγραμμάτων και των έργων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει ακόμη να συζητήσουμε και να βελτιώσουμε. Δημοσιονομικά μέσα. Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής έχουμε πάνω από χίλια δημοσιονομικά ε, νομοθετήματα. Τι είδους ε, ε, διαφάνεια λοιπόν είναι αυτή με την αντίστοιχη δημοσιονομική επιβάρυνση 900 εκατομμύρια ευρώ ε, διοικητικό κόστος με 6,7% των ε, πιστώσεων πληρωμών και ως εκ τούτου χαιρετίζω την πρωτοβουλία Κρέτσου και για μια πιο απλή και ολοκληρωμένη διαχείριση των κονδυλίων της περιφερειακής πολιτικής. Αυτά προς το παρόν από μένα σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. κυρία παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ, κύριε Σιγητά. Πιστεύω ότι καλύφθηκαν πολλά θέματα και προβλήματα και θα ήθελα να απαντήσω με τη σειρά. Πράγματι, η πολιτική συνοχή ορίζεται από την συνθήκη και νομίζω ότι έχει το στόχο να προσπαθήσει να μειώσει το χάσμα μεταξύ των περιφερειών αλλά και εντός των χωρών. Και σίγουρα τα ευρωπαϊκά ταμεία αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο. Όταν ε, μιλάμε για το ποσοστό σφάλματος για το 2016, γιατί αυτό συζητάμε σήμερα, τα κύρια είδη σφαλμάτων, όπως υπόθηκε εδώ ήταν ε, ε, κάποιες ε, παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, αλλά και κάποια μη επιλέξιμες δαπάνες και τα περισσότερα λάθη που ενιχνεύτηκαν από το ελεκτικό συνέδριο αναφέρεται σε λάθη που έχουν να κάνουν με την καταπάτηση της νομοθεσίας και των εθνικών κανονισμών. Γιατί μιλάμε για επιμερισμένη διαχείριση. Ουσιαστικά αυτά τα λάθη θα έπρεπε να ανακαλυφθούν από τις ε, διαχειριστικές αρχές που αποτελούν το πρώτο επίπεδο ελέγχου στις αντίστοιχες χώρες. Έτσι λοιπόν ε, τα προγράμματα και οι δικαιούχοι που δεν είναι επιλέξιμοι θα έπρεπε να έχουν ανοιχνευθεί κατά την επιλογή τους. Αυτό βέβαια μας ε, οδηγεί να σκεφτούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να βασιστούμε στις ελεγκτικές αρχές και εργαζόμαστε από κοινού όλα τα κράτη-μέλη για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στη διαχείριση σε ό,τι αφορά τις επαληθεύσεις που γίνεται στα διάφορα προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ανέφερε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος ε, των λαθών θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί από τις εθνικές αρχές που ελέγχουν τα προγράμματα βάσει των ε, πληροφοριών που είχαν. Έτσι λοιπόν, εμείς εκτιμάμε ότι το 72% των σφαλμάτων θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί αν οι εθνικές αρχές επεγρυπνούσαν περισσότερο και θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε αντί για 4,8% ε, ποσοστό λάθος, ε, για ποσοστό λάθος που να είναι κάτω από 1% πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη εποφελούνται από ένα εύρωστο σύστημα ελέγχου και παληθεύσεων. Και τότε Βεβαίως θα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτόν τον ενιαίο έλεγχο που είναι το όνειρο όλων των δικαιούχων και φυσικά είναι και προς όφελός μας. Πιστεύω ότι για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να σκεφτούμε την πολυπλοκότητα των κανονισμών, να σκεφτούμε αυτό το φαινόμενο του υπερθυματικού κανονισμού, της υπερβολικής νομοθεσίας ε, δηλαδή, το επίπεδο της συγκέντρωσης αλλά και την πιθανή έλλειψη εμπειρίας. Παραδείγματο χάρη σε πολλές χώρες έχουμε λάθη που οφείλονται στη διακύμανση ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του προσωπικού των διαχειριστικών αρχών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχώς παρακολουθούμε αν λειτουργούν καλά τα συστήματα και βασιζόμαστε στα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουμε στη διάθεσή μας. Χρησιμοποιούμε πλήρως ε, τα στοιχεία που έχουμε στις ετήσιες ε, εκθέσεις. Ε, λαμβάνουμε κατά μέσο όρο περίπου 500 εκθέσεις. Ο στόχος των ελεγκτών μας είναι τα προγράμματα μεγάλου κινδύνου Εκεί βλέπουμε ε, ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα προγράμματα στα κράτη-μέλη. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, έχει κάνει ε, πολλούς ελέγχους και τα δύο τρίτα αυτών των προγραμμάτων ε, διακόπηκαν μέχρι τη διόρθωση των σφαλμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ήδη έχουμε συμπεριλάβει νέα στοιχεία στον κανονισμό για την ετήσιο έλεγχο των προγραμμάτων στα συστήματα διαχείρισης και την ανείχνευση σοβαρών προβλημάτων εγκαίρως. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να βοηθούμε αλλά και να επιβλέπουμε τα κρατη Και φυσικά εκεί όπου βλέπουμε μεγάλες αδυναμίες δηλαδή αντίκτυπο πάνω του 10% στα μετά με τις πληρωμές. Σε σχέση τώρα με τις καθυστερήσεις, τις οποίες αναφερθήκατε, είναι κάτι που μας ανησυχεί. Ταυτόχρονα χαίρομαι που βλέπω μία επιτάχυνση ε, στην εφαρμογή αν ε, είχα έρθει πριν μία εβδομάδα στην Κέση Επιτροπή, θα είχα μιλήσει για 30% ε, ε, στο επίπεδο επιλογής και μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε φτάσει τώρα στο 40% σε επίπεδο κρατών μελών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εφαρμογής στις κάτω χώρες όμως αυτό, παραδείγματο χάρη, δεν μεταμορφώνεται σε αιτήσει πληρωμής προς την Κομισιόν, γιατί ήδη έχουν λάβει τις προκαταβολές, ήδη έχουμε εκεί ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και έχουμε ε, στείλει σε πολλά κράτη-μέλη ε, τίματα από τους τέσσερις επιτρόπους για την επιτάχυνση των ε, πληρωμών. Έχει γίνει η εφαρμογή, έχει γίνει και η επιλογή, όμως παρόλα αυτά δεν έχουμε αιτήματα πληρωμής από τις κάτω χώρες. Και άλλα κράτη-μέλη τα πάνε πολύ άσχημα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και δεν έχουν λογαριασμούς να μας στείλουν. Η απλούστευση λοιπόν αποτελεί η μέγιστη προτεραιότητα για μένα. Είμαι πεπισμένη ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική που ε, εδώ και 20 χρόνια δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει μεταρρυθμιστεί, εδώ και 25 χρόνια έχουμε την πρόταση της Κομισιόν, το Omnibus, στην οποία προστίθεται πάνω από χίλιες τροποποίησεις εγώ βασίζομαι στην ε, δική σας υποστήριξη αυτό που θα βγει από το Omnibus ε, να μην είναι πιο πολύπλοκο από αυτό που προτείνουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των δικαιούχων ε, και να γίνει πιο εύκολη η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τώρα, σε σχέση με τον νέο έλεγχο. Έχουμε επισκεφτεί πολλά κρατημέλη, δεκάδες περιφέρειες που λαμβάνουν ε, ουσιαστικά τα ίδια ε, παραπάνω. Παραδείγματο χάρη στην Ανατολική Γερμανία, οι περισσότερε μικρέ και μακρισέ επιχειρήσει αποτελούνται από 5-6 ανθρώπου ε, και κάποια μέρα πάνε 80 άνθρωποι να του κάνουν έλεγχο μέσα σε μόνο και μία μέρα. Σίγουρα το επόμενο έτος αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Κάτι τέτοιο πρέπει να το αποφύγουμε. Σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, πιστεύουμε ότι αυτή η διεύρυνση ε, έχει βοηθήσει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο ήδη αυτά τα μέσα. Υπάρχουν και κάποιες καινοτομίε για την περίοδο 2007-2013. Για την περίοδο 2014-2020 έχουμε διπλή πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά μέσα, γιατί αυτά αποτελούν πολύ αποτελεσματικό τρόπο ενεργοποίησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την επίτευξη των στόχων αναχώρα αλλά και των στόχων μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε ε, κάποια παραδείγματα των πρακτικών. Μπορούμε να τα βασίσουμε ε, στις εμπειρίες που έχουμε και ελπίζω ότι με το νέο νομικό πλαίσιο και με την ε, ικανότητα που θα μας δώσει το Omnibus να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τον ε, αντίκτυπο των χρηματοοικονομικών μέσων ε, γιατί πράγματι αυτά πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχουν κίνδυνοι και συμβαδίζουν ε, με ε, τις επιδοτήσεις. Από την άλλη, η υιοθέτηση του Omnibus θα καταστήσει δυνατή και την συμπληρωματικότητα μεταξύ των διορθωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Ταμείου του σχεδίου Juncker δηλαδή. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποια από τις ερωτήσεις σας. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι βάζουμε τα δυνατά μας για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Σε σχέση με το ΕΦΣΥ, μιλάμε για 315 δισεκατομμύρια πέρα από τα δικά μας κονδύλια μέσω του Omnibus ε, προσπαθήσαμε να έχουμε μια συνδυασμένη χρηματοδότηση που να είναι πιο δυνατή, χρησιμοποιώντας και μια κοινή πλατφόρμα επενδύσεων στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη-μέλη. Και αναφερθήκατε και σε κάποιες προκαταβολές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ε, πληρωμές που έχουν κίνδυνο. Το ελεκτικό συνέδριο Αναφέρθηκε σε κάποια μεθοδολογικά σημεία σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά μέσα. Σας διαβεβαιώ ότι συνεργαζόμαστε με το Ελεκτικό Συνέδριο και με τα κράτη-μέλη για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να βρούμε μία λύση στην προβληματική που θέσατε. Όμως, όπως είπατε και εσείς, είμαι πεπισμένη ότι από κοινού μπορούμε να εργαστούμε και να συνεργαστούμε και με το Ελεκτικό Συνέδριο που έχει πολύ ανοιχτό πνεύμα για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των Ευρωπαϊκών Ταμείων και να βασιστούμε περισσότερο και στις ελεγκτικές αρχές, γιατί αυτό είναι βασική προϋπόθεση για την απλούστευση και για να έχουμε καλύτερη διαχείριση. Είναι πολύ λυπηρό κατά την άποψή μου να βλέπει κανείς ότι το 7% των λαθών δεν έχουν ε, εντοπιστεί εκεί που θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί και θα έπρεπε να έχουμε τον έλεγχο της ΟΛΑΦΗ του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Κομισιόν ε, για να εντοπίσουν τα λάθη αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ είναι η επόμενη στον ε, κατάλογο. Ας σας ελέγξουμε πρώτα μερικά ερωτήματα. Σας ακούμε. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, καθώς ε, βλέπουμε ότι αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη ταχύτητα και εμφανίζονται και κάποια σημεία εμπλοκής που θα πρέπει να εξαλείψουμε για το μέλλον. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εντός των δύο συστημάτων του τρόπου χρηματοδότησης, πέρα από το καινοτόμα εργαλεία. Αλλά όταν μιλάμε για τα κονδύλια που δίνονται σε περιφερειακό επίπεδο από την πρώτη μέρα της ε, συμφωνίας του Συμβουλίου για την κατανομή και τα κονδύλια που επιτυγχάνονται μέσω του, ρίζετος ε, του, του προγραμμάτος 2020 και ε, άλλων τρόπων. Θέλω να σας ρωτήσω την εμπειρία που είχατε. Δηλαδή, ακούγεται όλο ένα και περισσότερο για το μέλλον ότι αν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, περιοριστεί, να υπάρξει η δυνατότητα να απαιτηθεί τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία να μπουν περισσότερο σε αυτή την άλλη φόρμουλα σχεδίων που θα χρηματοδοτούνται μέσω ε, κάποιων ε, τρόπων δημοπρασίας. Θα ήθελα να μου πείτε, αν από την εμπειρία που έχετε και φυσικά έχοντα και κατά νου το πώ θα γίνει ο έλεγχο, αν μπορεί να γίνει ένα μείγμα μια ε, κατανομή. Να υπάρχει δηλαδή ε, ουσιαστικά και το πόνους μέσα από τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα, για να υπάρχει κάποιο κίνδυνο και για το χρονοδιάγραμμα. Εμείς ε, ξέρουμε ότι στο τελευταίο οικονομικό έτος η καθυστέρηση οφειλόταν ε, στην ε, καθυστερημένη υιοθέτηση, στο ότι άργησαν οι να προσαρμοστούν ε, στο νέο στη νέα προγραμματική περίοδο για το μέλλον. Ο κύριος Έτικερ θα παρουσιάσει την πρόταση το Μάιο-Ιούνιο του 2018. Θα μας μείνει μόνο ένα χρόνο, ένας χρόνος σε εμάς το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να το υιοθετήσουμε και η Κομισιόν θα έχει λίγους μήνες ακόμα για να το θέσει σε εφαρμογή πριν από την ε, έλευση της νέας Κομισιόν. Έτσι λοιπόν πώς βλέπετε εσείς αυτό το χρονοδιάγραμμα, τι εμπειρίες έχετε από τις ε, καθυστερήσεις, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το επόμενο οικονομικό έτος ε, και να δούμε και τι θα γίνει και με το Brexit παραλλήλως. Και τέλος, ξέρετε ότι και εμείς και η Κομισιόν αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα για μεγαλύτερο ποσοστό ευελιξίας. Δηλαδή να μην ε, έχουμε άμεση ε, κατανομή του προϋπολογισμού. Πώς βλέπετε εσείς ότι αυτή η ευελιξία θα μπορούσε να μας βοηθήσει έτσι ώστε τα διαφορετικά ταμεία να είναι λιγότερο μακροπρόθεσμα. Γιατί έχουμε τώρα εδώ όλες αυτές τις καθυστερήσεις, ε, τα λανθασμένα project, τις απαραίτητες διορθώσεις κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει την πολιτική συνοχή να υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία και ένας μεγαλύτερος ρεολισμός ως προς την προσαρμογή το σύστημα των ε, καθαρών, ε, των καταποκοπή διορθώσεων, που στους περισσότερους εδώ στο Κοινοβούλιο φαινόταν ένα πιο αυστηρό ή πιο αποτελεσματικό σύστημα για να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να μην διαπράττουν σφάλματα. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη, επειδή φοβούνται αυτές τις διορθώσεις, βλέπουμε ότι καθυστερούν, χρονοτριβούν. Ακριβώ επειδή φοβούνται αυτές τις ε, καθαρές διορθώσεις. Έτσι λοιπόν, ένα εργαλείο που φαινόταν καλό, τελικά καταλήγει να είναι ένα εργαλείο το οποίο επιφέρει προβλήματα. Θα ήθελα τη γνώμη σα από αυτού. Κυρία Χλαμπάγιο, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ξέρετε κύριε Επίτροπε ότι υποστηρίζω την πολιτική συνοχής ιδιαίτερα και τον προϋπολογισμό με βάση τα αποτελέσματα και την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία στα προγράμματα. Επιτρέψτε μου όμως ε, να διατυπώσω με διαφορετικές προοπτικές αυτή τη φορά τα ερωτηματικά μου. Το 2016 ήταν το τελευταίο έτος της ε, επαλήθευσης εκτέλεσης του προπολογισμού του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2017-2016 2013-2017 με ε, την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρχει ε, υπολοιπόμενος κίνδυνος για την εκτέλεση. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν, η Επιτροπή βλέπει κάποιο πρόβλημα σε ολοκλήρωση κλείσιμο συγκεκριμένα προγραμμάτων και στις διαδικασίες των διορισμών που μας ανέφερε και ο εισηγητής μας. Θα μπορούσε ε, μια λύση να ήταν αντί για αποτελέσματα και αντίκτυπο για τον ε, πολίτη να κατηγορηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ακόμα στις δομές δείχνει τα χρήματά της και σύμφωνα με, τον κύριο, με τα όσα είπε και ο κύριος Τσέλερ θέλω να ρωτήσω τεχνογνωσία, υπηρεσίες συμβουλών ε, είναι απαραίτητες το κόστος που έχουν στον προϋπολογισμό ύστερα από τρία χρόνια λειτουργίας της πολιτούς δημοσιονομικής περίοδου. Είναι τόσο περίπλοκος ο κανονισμός. Είναι τέτοιες οι αποτυχίες των κρατών μελών και τα δύο. Επίσης, κυρία Επιτροπέ, σε σχέση με το πρόγραμμα δράσεως για τις δημόσιες προμήθειες του 2013, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2015 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πρόσθετα προληπτικά μέτρα, καθοδήγηση, κατάρτιση, βέλτιστες πρακτικές, ε, κατάλογος των ε, προς αποφυγή λαθών και το καθεξής. Επικαιροποιήθηκε το Μάρτιο του 2017 μάλιστα, μόνο όμως τότε, για να συμπεριλάβει και τις ατάξεις που προκύπτουν μετά την ε, νέα οδηγία και τις προτάσεις και διατάξεις για τη διαφάνεια. Ε, οι οδηγίες λοιπόν που υιοθετήθηκαν το 2014 για τις δημόσιες προμήθειες και αναφέρονταν σε νέες δράσεις και ζητήματα ε, μεταφοράς. Όταν η μεταφορά γίνεται το 2017 δεν είναι αργά και άμα λάβουμε υπόψη και το πόσο τα κράτη-μέλη προσαρμόζουν προς όφελός τους τις οδηγίες αφενός. Αφετέρου δεν τις καθυστερήσεις στο επίπεδο επιτροπής δεν θα ήταν λιγότερο δαπανηρό αλλά και πιο αποτελεσματικό να έχουμε κανονισμό αντί για οδηγία ως ε, νομοθετική πράξη. Τι λέτε εσείς και τι θα έλεγε και το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στη διαδικασία της απαλλαγής. Ναι, και εγώ έχω βάλει το όνομά μου στον κατάλογο των αγορητών. Για τον ε, χάρτη. Αυτόν είναι η ερώτησή μου που αναφέρεται στις διαδικασίες των ε, προμηθειών και διαρωτώ με πώς είναι τόσες οι περιφέρειες και δει στην Ελλάδα, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ιταλία να έχει κερδίσει την πλειοδοσία ένας και γιατί καμία άλλη επιχείρηση δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Τι κάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. Τι είναι αυτές οι, αυτές οι προμήθειες, είναι η γαλακτοφόρος, η χρυσοφόρος μάλλον αγελάδα των τραπεζών από τα δημοσιονομικά μέσα. Εδώ έχουμε 900 εκατομμύρια. Είναι χρήμα το οποίο τελικά θα λείψει από κάπου αλλού, από τον κορβανά μας. Στην αρχή τα απορροφούσαν τα κράτη. Ε, τώρα πάνε στις τράπεζες. Με τι αποτέλεσμα στην ερώτηση δε 67 λέτε ότι το διαχειριστικό κόστος είναι 2,6% αναέτος. Δηλαδή 5,3 συνολικά. Ε, μάλλον όχι. Έχετε υπολογισμό 5,3 έτη. Γιατί όχι 7 στο δημοσιονομικό μέσον. Το 5,3 δεν το καταλαβαίνω. Και ίσως θα πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί εξακολουθείτε να ανέχεστε την ε, στάθμευση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών μέσων. Πρέπει να ρίξουμε μια ματιά πιο προσεκτική στην ερώτηση 57. Η ερώτηση νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα από την απάντηση. 170.000 θέσεις εργασίας λέτε. 680 θέσεις ανά κράτος στατιστικά, αν κάνουμε έναν επιμερισμό. Δεν φαίνεται δηλαδή ε, τα δημοσιονομικά μέσα που διαθέτουμε να ε, στέφονται και με φοβερή επιτυχία ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πώς θα κρίνετε λοιπόν εσείς αυτά τα δημοσιονομικά μέσα και τι θα γίνει από εδώ και μπρο. Στην προσεχή δημοσιονομική περίοδο και τέταρτη ερώτηση. Το ελεγκτικό συνέδριο στο 6-19 λέει ότι έχει 3,7% ποσοστό λάθος, το χαμηλότερο σε, διαχειριστικές, ε, σε αρχές διαχειριστικές. Ε, όμως ένα single audit ίσως, και δεν το κοιτάει κανείς αυτό, οι διαχειριστικές αρχές μας δίνουν στοιχεία με πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Είναι αποδεκτό το ποσοστό αυτό, βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο δηλαδή, δεν το ανασκάπτουμε, δεν το ψάχνουμε περισσότερο. Κύριο Αλαφράγκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που είναι σήμερα εδώ και απαντά στις ερωτήσεις των βουλευτών. Και ευχαριστούμε και για το ερωτηματολόγιο η πρόεδρος της Επιτροπής μας ε, έκανε την ερώτηση που ήθελα να κάνω κι εγώ. Γιατί και μένα μου τράβηξε την προσοχή το γεγονός ε, ότι στη διαχείριση των 35 ε, δισεκατομμυρίων στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής πέρσι το ποσοστό λάθους ήταν 4,8% και μας λέει ότι αν οι εθνικές αρχές είχαν εφαρμόσει σωστά τους μηχανισμούς ελέγχου, αυτό αυτό το ποσοστό θα ήταν στο 1,1%, δηλαδή κάτω του 2%. Μιλάμε εδώ για προγράμματα χρηματοδότηση όπου οι εθνικέ αρχέ επίση έχουν ε, ευθύνη στη διαχείριση. Υπάρχουν ε, όμω και άλλα στοιχεία, υπάρχει άλλο ένα στοιχείο και θα σα ρωτήσω κύριε Επίτροπε, στην έκθεση του Νεκτικού Συνεδρίου λέγεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν διορίσει μόνο το 75% των εθνικών αρχών αρμοδίων ε, για την εφαρμογή των αντίστοιχων κονδυλίων. Δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί αυτό το νούμερο και αν η Κομισιόν ε, γνωρίζει αυτή την ε, πληροφορία. Γιατί τρία έτη μετά από τη θέση σε ισχύ των δημοσιονομικών προοπτικών, ακόμη να μην έχουν διοριστεί 100% οι εθνικέ αρχέ για την εφαρμογή των κονδυλίων, νομίζω ότι αυτό εξηγεί πολλά μεταξύ άλλων σε σχέση με τι σημαντικέ καθυστερήσει που βιώνουμε. Κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν ε, με την επίτευξη των στόχων αυτών των πολιτικών και συγκεκριμένα σε τρεις κυρίες πτυχέ. Στην προσθέμενη αξία αναφέρθηκε συνάδελφος, είναι σημαντικό κριτήριο. Το δεύτερο, σε ποιο βαθμό η χρήση των κονδυλίων μπορεί να συνεισφέρει στην καινοτομία που είναι θεμελιώδης παράγοντας ανάπτυξης. Ε, εγώ καταλαβαίνω ότι ε, δεν μπορούν να είναι όλοι πρωτοπόροι ε, σε αυτό το επίπεδο, αλλά η καινοτομία είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σας θέσω και δύο σύντομες ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ποιο βαθμό η μεταναστευτική πίεση που βίωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε συνέπειες ε, στην διαχείριση των διαφορετικών ταμείων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο αυτό και να μας πείτε αν κατά τη γνώμη σας έχουμε επαρκή εργαλεία για να ε, επιλύσουμε ευέλικτα αυτό το πρόβλημα. Και κάτι ακόμη, διάβασα τα στοιχεία από τις απάτες ε, που έχουν λάβει η χώρα και σύμφωνα με την έκθεση του Λεκτικού συνεδρίου είναι μειωμένα. Πώς εργάζεστε εσείς ε, με την ε, Όλαφ, πώς συνεργάζεστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Ελληνικού Συνεδρίου, τρίτη φορά ακούω το ποσοστό λάθους και μου έρχεται να βάλω τα γέλια. Τι είναι το ποσοστό λάθους. Αν δούμε τη σύγκριση μεταξύ των διαφορών κρατών μελών, εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει χαμηλότερο ποσοστό λάθος στην Ελλάδα από ό,τι στην Τσεχία. Αλλά εκεί δεν χρησιμοποιείται και η ίδια μέθοδος. Μπορεί λοιπόν σε ένα κράτος μέλος το ποσοστό λάθος να είναι πιο υψηλό και σε άλλο πιο χαμηλό. Έχω ξαναπεί ότι πραγματικά δεν είναι σημαντικό αυτό για, τον, για τους ελέγχους αν έχω λάθη ή αν έχουν δηλωθεί τα λάθη ή όχι. Η κυρία Επίτροπε, είπατε ότι οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουν να χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ πριν ε, γίνω μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δούλεψα σε τέτοιε εταιρείε και πραγματικά ποτέ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιώ ευρωπαϊκέ ενισχύσει γιατί η γραφειοκρατία είναι τραγική. Και τα τελευταία τρία χρόνια, όποτε επισκέπτομαι επιχειρήσεις, βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε. Ίσως ε, εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρείτε ότι ε, έχετε προχωρήσει ουσιαστικά, αλλά έχουμε 40 έγγραφα για να μπορέσουμε να, κάνουμε, να υποβάλουμε μια αίτηση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να το κάνουμε από το ίντερνετ. Αντί να πρέπει να κατεβάζουμε δεκάδες έγγραφα. Ως προς αυτό λοιπόν, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή έχει μεγάλη δουλειά να κάνει και δεν νομίζω ότι έχετε καταφέρει πολλά. Δεύτερον, ε, Κομισιόν απέναντι στα κράτη-μέλη. οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι για την ε, τυπογραφία στην... Ε, έχουν καταστρέψει την τυπογραφία στην ε, Τσεχία. Οι συνθήκες εργασίας γίνονται χειρότερες στην βιομηχανία αυτή. Όλο και λιγότεροι εργάζονται στην βιομηχανία αυτή και ποιο είναι το αποτέλεσμα τελικά τι έπρεπε να έχουμε πετύχει με αυτές τις επιδοτήσεις. Ουσιαστικά τα χρήματα αυτά τελικά επενδύονται σε ανοησίες. Και ένα τρίτο ερώτημα για την απορρόφηση των κονδυλίων. Ε, είπαμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν τα συγκεκριμένα κονδύλια. Για το 2018 δεν θα πρέπει κάτι να αλλάξει. Πότε θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ξεκινούν με την απορρόφηση των κονδυλίων. Ε, δεν κατάλαβα τι ακριβώς ήταν η βιομηχανία στην οποία αναφερθήκατε και το έψαχνα κιόλας. Ο συνάδελφος Βόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που άργησα να έρθω και ελπίζω να μην, να πρόκειται να πω κάτι που το έχετε ήδη πει. Ευχαριστώ την ε, ε, πίτροπο που ε, είναι σήμερα εδώ. Είναι γνωστή φυσιογνωμία στην Επιτροπή. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Σαλαφράγκα για τις περιπτώσεις απάτης οι απάτες είναι, αρκετά χαμηλές και λυπάμαι που μερικοί συγχέουν τις απάτες με τα λάθη. Τα λάθη, τα σφάλματα είναι κάτι διαφορετικό και κάθε ευκαιρία που έχουμε αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Υπάρχει διαφορά μεταξύ απάτης έτσι ώστε οι ευρωσκεπτικιστές να μην μπορούν να λένε ό,τι θέλουν σχετικά. Βεβαίω πρέπει να μειωθεί το ποσοστό λάθους, βεβαίω έχουμε κάνει πολλέ συζητήσει από αυτού στο παρελθόν, βεβαίω υπάρχει ανάγκη για απλούστευση, έχουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση και η επίτροπο λέει ότι οι συστάσει που υπάρχουν από το ελεκτικό συνέδριο θα κάνουν τη διαφορά σε ό,τι αφορά την απλοποίηση των πραγμάτων και τη μείωση του ποσοστού λάθου. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και για τα κράτη-μέλη και για αυτόν τον υπερθεματισμό σε ό,τι αφορά την ε, νομοθεσία. Ελπίζω ότι, αυτό που θα κάνουμε είναι να ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα και να... μην το συζητούμε χρονιά τη χρονιά, αλλά να βρίσκουμε τελικά τη λύση του έτσι ώστε στο τέλος να κάνουμε αυτό που ε, είχαμε βάλει ως στόχο, να μειώσουμε δηλαδή το λάθος. Τώρα, για, τις, ε, για το ποσοστό απορρόφησης, ξέρουμε ότι τα κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό απορρόφησης Παρ' όλα αυτά υπάρχει γενικό ποσοστό απορρόφηση 70%, τα πάμε αρκετά καλά λοιπόν. Βεβαίω τώρα είμαστε στον κανόνα νήσιν 3, οπότε αυτό το έτος είναι πολύ σημαντικό. Ερώτημα λοιπόν ως προς αυτό. Είναι δυνατόν, είναι πιθανό τα κράτη-μέλη να ε, σταματήσουν να χρησιμοποιούν κάποια κονδύλια ακριβώ λόγω της χαμηλής απορρόφησης που έχουν και για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα που είναι αρκετά αντιφατικό θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία απειλούνται από αυτό. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο λοιπόν να το δουλέψουμε. Ερώτημα, είναι δυνατόν στο μέλλον να απομακρυνθούμε από αυτό και να μην πιέζουμε τα κράτη-μέλη τόσο πολύ, αλλά να μιλούμε κυρίως για τα project και τις περιφέρειες που θα τα διαχειριστούν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να χαιρετήσουμε και τον Γενικό Διευθυντή, δεν ήθελα να το ξεχάσω. Ε, κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Αναφέρθηκαν ε, πολλά θέματα. Να ξεκινήσω από μια διαπίστωση. Δυστυχώς βλέπω ότι όλο ένα και περισσότεροι βουλευτές ε, μιλούν ε, από την αρχή για μειωμένο προπολογισμό. Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Ο κύριος συζητητής, ο κύριος Τσέλερ, μίλησε για τις δηλώσεις ε, του πρόεδρου Γιούνκερ, καθώς και του Επιτρόπου Έτινκερ, που είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια συζήτηση για το μελλοντικό ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση αυτή και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη με αφετηρία τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και βρίσκοντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ των πολιτικών που λειτουργούν, των πολιτικών που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στη ζωή των πολιτών και τις ε, νέες προτεραιότητες ε, άμυνα, μετανάστευση, έλεγχο των συνόρων καθώς πρόκειται για τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα δεν είχε αρμοδιότητε ε, ή μόνο πολύ μικρέ αρμοδιότητε. Θα υπάρχουν και άλλε ε, συζητήσεις εδώ για το σε ποιο βαθμό θα συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμεσα, έμεσα ή μέσω τη επιμερισμένη διαχείριση. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία περιφέρεια πλούσια φτωχή που να μην έχει δει αυτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία μου δίνουν ε, ενέργεια να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την περιφερειακή πολιτική, γιατί ξέρουμε ότι χάρη σε αυτές τις περιφερειακές πολιτικές έχουν δημιουργηθεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας, και ακόμη και τα κράτη-μέλη που είναι καθαροί συνεισφέροντες έχουν επωφεληθεί από την αύξηση του εμπορίου. Μετά από τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα δούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα περιορισμένο προϋπολογισμό ή για έναν προϋπολογισμό που να αποτελεί το 1% του ακαθαρίστου εγχώριου εισοδήματος, ε, κατά κεφαλήν εισόδημα για τα 27 κράτη-μέλη στο μέλλον, το 2020, ή αν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα φιλόδοξο επίπεδο, δηλαδή στο 1,2% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος των 27 κρατών μελών για να διατηρήσουμε τις πολιτικές που έχουν αποδειχθεί ωφέλιμες για τους πολίτες. Ταυτόχρονα μπορέσουμε να εισαγάγουμε και νέες προτεραιότητες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει για να απαντήσει στις νέες προκλήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό σημαίνει η ελληνική, το να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τα κράτη-μέλη και να δούμε αν είναι διατεθειμένα. Σίγουρα εμείς θα πρέπει να απλωστεύσουμε, να μειώσουμε και να εξαλείψουμε τις ε, επικαλύψεις Υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, συγκρούσεις ε, μεταξύ των διάφορων κανονισμών. Όμως πρέπει να ρωτήσουμε και τα κράτη-μέλη αν είναι διτεθειμένα να συνεισφέρουν περισσότερο ή αν θέλουν να εγκαταλείψουν αυτές τις πολιτικές. Για κάθε 100 ευρώ που δίνει ο καθένας σας, τα 50 πάνε σε φόρους και στην ασφάλιση και λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα πηγαίνει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δηλαδή, εμείς ε, για ε, ένα ποσό που αντιστοιχεί σε ένα καφέ ή σε ένα μπουκάλι νερό, καλούμαστε να συνεισφέρουμε στην κοινή αγροτική πολιτική, στην πολιτική συνοχή, στην έρευνα, στην καινοτομία και στις υπόλοιπες προτεραιότητες. Σίγουρα, εγώ δεν θέλω τώρα εδώ να προκρίνω, όμως πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, πιστεύω. και να μην ε, αναφέρουμε κάτι ως δεδομένο. Ναι, εντάξει, θα έχουμε τον Brexit, αλήθεια είναι, αλλά να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Έχουμε και την έκθεση Μόντι για να αυξήσουμε τα έσοδα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και να δούμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη θα δεχτούν τις προτάσεις αυτές. Αυτή είναι μια πολιτική παρατήρηση που σχετίζονται με αυτή την έκφραση που ακούω όλο ένα και πιο συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ υπάρχει μια απεσιοδοξία για έναν περιορισμένο προπολογισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γιάλα. Συμφωνώ μαζί σας. Πρόκειται για ένα πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Ο πρόεδρος Γιούνκερ, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι το σχέδιο προπολογισμού θα κατατεθεί το Μάιο. Εμείς ελπίζουμε ότι οι κανονισμοί για την ε, περίοδο μετά το 2020 να ακολουθήσουν αμέσως και ελπίζουμε να έχουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε και από τη δική σας θητεία να υλοποιηθούν αυτοί οι κανονισμοί γιατί ουσιαστικά οι κανονισμοί γίνονται από το προηγούμενο κοινοβούλιο και ο προεπλογισμός έχει χτιστεί από το προηγούμενο κοινοβούλιο και είναι κρίμα η δική σας εμπειρία να μην συνεισφέρει στους κανονισμούς μετά το 2020. Σε σχέση τώρα με την ευελιξία στην οποία αναφερθήκατε, δεν μπορούμε να προκρίνουμε είναι βέβαια ένα θέμα που βρίσκεται επιτάπητος, να είμαστε δηλαδή πολύ πιο ευέλικτοι σε θέματα όπως είναι η μετανάστευση, φυσικές καταστροφές και άλλα ζητήματα, όπου θα πρέπει να αντιδρούμε πιο γρήγορα και να βοηθάμε τα κράτη-μέλη. Σε σχέση τώρα με τις κατακοπήν διορθώσεις. Υπάρχουν ε, πολύ σωρευτικοί παράγοντες και το γεγονό ότι άργησε να θετηθεί το πολιτεστικό συνομικο πλαίσιο και ότι είχαμε αυτόν τον κανόνα νήσιν 3 που κάπως ε, χαλάρωσε την πίεση στα κράτη-μέλη. Και ο τρίτος λόγος είναι ο φόβος ε, απέναντι σε αυτές τις διορθώσεις. Ε, αυτός ο φόβος μας διαβεβαιώνει ότι έχουμε ελέγχους ποιότητας, για να το δούμε θετικά, και είμαστε σίγουροι πως όταν λαμβάνουμε αυτούς τους ελέγχους, αυτή είναι ποιοτική, Ελπίζουμε ότι με την εισαγωγή αυτών των καθαρών διορθώσεων οι διαχειριστικές αρχές, όπως είπαμε, θα πρέπει να είναι το πρώτο επίπεδο ελέγχου ε, να γίνονται λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι σε αυτό το επίπεδο με μεγαλύτερη ε, αυστηρότητα και με καλύτερο τρόπο για την περίοδο μετά το 2020. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η περίοδος αυτή. Χρειαζόμαστε μια ανάλυση για το πώς εφαρμόζεται ο προπολογισμό επιτόπου. Όπως είπα, χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία εγώ είμαι υπέρ μιας ριζικής απλούστευσης για τους δικαιούχους αφενός και αφετέρου πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε και σε θετικά στοιχεία του σημερινού συστήματος. Να βρούμε δηλαδή τη σωστή ισορροπία μεταξύ της μεταρρύθμισης και της συνέχειας. Και εδώ θέλω να φερθώ και στο τύπο κύριο Βόγκαν, γιατί τα λάθη δεν σημαίνουν απάτες. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τη συνολική εικόνα της πολιτικής συνοχής σε όλα τα κράτη-μέλη. Από την άλλη, θα πρέπει βέβαια να παρεμβαίνουμε εκεί όπου υπάρχουν αδυναμίες. Σε σχέση με το στάδιο του κλεισίματος του προγράμματος 2007-2013, ε, αυτό που ρώτησε η κυρία Ντεμπέβλα και την ευχαριστώ για τη συνεργασία μας όταν ήσασταν συγγήτρια. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή ε, έχει γνωμοδοτήσει θετικά για το κλείσιμο της περίοδου 2007-2013. Δημοσιεύτηκε και μια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου σε σχέση με το επίπεδο προετοιμασίας μας για το κλείσιμο του προγράμματος και γενικά ήταν θετικό το αποτέλεσμα. Οι οδηγίες της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη ήταν πλήρες και δόθηκαν εγκαίρως μπορώ να πω ότι όλα τα έγγραφα που αφορούν το κλείσιμο ελήφθησαν εγκαίρως, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο του 2017. Ξέρετε ότι αυτή ήταν η καταληκτική προθεσμία κλεισίματος για το πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και από 400 συμπρογράμματα προγράμματα που είχαμε στα 28 κρατημέλη. Οι υπηρεσίες μας έστειλαν τις αξιολογήσεις ε, στα κράτη-μέλη μέσα στην προθεσμία. Τώρα έχουμε κλείσει μόνο 9 προγράμματα από 417. Γιατί ζητήσαμε και πρόσθετες πληροφορίες εκεί όπου χρειαζόταν. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να κλείσουμε από 80 έως 120 μέχρι τα τέλη του 2017 αναμένοντας ε, να λάβουμε και τις πληροφορίες που έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη. Έχουμε βέβαια και κάποια αιτήματα που δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουμε ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις ή πρόσθετες επαληθεύσεις, απαραίτητες ε, οικονομικές διορθώσεις. Κάποια κράτη δέχονται, κάποια κράτη δεν δέχονται αυτές τις διορθώσεις, ότι όλα αυτά τα προγράμματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι ότου όλα τα αιτήματα να υλοποιηθούν. Εν τω μεταξύ, εμεί κάνουμε διάμεσε πληρωμέ για τα προγράμματα που θεωρούνται σίγουρα. Δηλαδή, ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει σε ένα πρόγραμμα που το θεωρούμε επικίνδυνο. Δεσμευόμαστε, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στο να κλείσουμε τα προγράμματα το συντομότερο. Από την άλλη όμως, όπως και στην περίπτωση της προετοιμασίας των προγραμμάτων, προτιμάμε να έχουμε μια ποιοτική διαδικασία για ε, το ένα ε, ποσοστό πληρωμών το 2% και σας είπα ότι θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει λάθος σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί. Τα κράτη-μέλη έχουν αναφέρει ένα υπολοιπόμενο κίνδυνο κατά μέσο όρο 2%. Όμως νομίζω ότι αργότερα θα μπορέσουμε να σας ε, παρουσιάσουμε και άλλα στοιχεία εδώ στο Κοινοβούλιο ως προς τα αποτελέσματα του κλεισίματος. Αυτό θα γίνει στις επόμενες ε, εκθέσεις δραστηριοτήτων. Για την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε και γραπτός έχω λάβει αυτή την ερώτηση και εμείς αναρωτιόμαστε για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μόνο έναν πλειοδότη ο οποίος ε, γράφεται σε μία και μόνο εταιρεία και μαζί με τον ε, Γενικό Διευθυντή ξεκινήσαμε μία έρευνα για τις περιπτώσεις αυτές στις οποίες εσείς αναφερθήκατε, κυρία Πρόεδρε. Έχετε δίκιο, πιστεύω. Πρέπει να μας απασχολούν τα θέματα αυτά, έχουμε ερωτηματικά καθώς ε, είναι και ε, πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός ε, σε ό,τι αφορά την απόκτηση κάποιων σχεδίων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων, όπως είπα, χρησιμοποιήθηκαν ήδη από την περίοδο 2000-2006, διαδόθηκαν περισσότερο στην περίοδο 2007-2013, όμως βλέπουμε ότι είχαμε σημαντικά αποτελέσματα επιτόπου. Ξέρω ότι εσείς αναφέρεστε στις ε, στις 17.000 θέσεις ε, που δημιουργούνται στα κράτη-μέλη κάθε χρόνο. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι απολύτως πλήρη Είμαι πεπισμένη ότι θα υπάρχει πολλαπλασιασμός ε, αυτών των θέσεων εργασίας σε την ακόλουθη περίοδο. Σας ε, έχω απαντήσει γραπτός στην ερώτηση 75. Ξέρετε ότι στην περίοδο 2007-2013 τα κράτη-μέλη δεν υποχρεώθηκαν να μας δώσουν αυτούς τους δείκτες. Εμείς ε, δίνουμε αυτά τα στοιχεία βάσει δικτών που μας έδωσαν κάποια, πρακτι... κάποια κράτη-μέλη εθελοντικά. Για την περίοδο όμως 2014-2020 θα υποχρεωθούν να μας δώσουν λεπτομερώς αυτούς τους δείκτες. Έτσι λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα στοιχεία. Πιστεύω ότι τα δικά μας δεδομένα δείχνουν ότι συνολικά επενδύθηκαν 17,4 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοοικονομικά μέσα, 89% σε ό,τι αφορά την βοήθεια σε μικρές και μεσές επιχειρήσεις, 4% σε ενεργειακή αποδοτικότητα και 13.500 τελικοί δικαιούχοι υποφελήθηκαν από αυτά τα ταμεία και δημιουργήθηκαν 170.000 θέσεις εργασίας. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η μόχλευση είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε κάποιες χώρες όπου σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουμε σε πάνω από 20 φορές μεγαλύτερη μόχλευση για τις εγγυήσεις ε, και για τα δάνεια. Στην Αυστρία και στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, αυτέ είναι οι χώρε που υποφελούνται από κονδύλια από το σχέδιο Μάρσελ, λόγω αυτού του αποτελέσματος της μόχλευσης, αυτού του φαινομένου της μόχλευσης. Πιστεύω ότι η διοικητική ικανότητα των χωρών αυτών να χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά εργαλεία και να μεγιστοποιούν την δυνατότητα χρήσης τους. Σε σχέση τώρα με την ερώτηση του κυρίου Σαλαφράνκα. Όπως σας είπα, κύριε Σαλαφράνκα. δεν υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον διορισμό, τον καθορισμό των αρχών καλύπτουμε τώρα το 98% ε, σε ό,τι αφορά τα ταμεία συνοχής και τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης. Βέβαια πρέπει να γίνουν κάποιοι διορισμοί σε ό,τι αφορά τον τομέα της ε, εδαφικής συνεργασίας, όμως γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι αυτή η καθυστέρηση οφείλεται και στο γεγονό των πολυπλοκοτήτων της εξάντερης ε, που είχαμε σε σχέση με τις συστάσεις ένα χώρα. Αυτό μας βοηθά να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι φορείς θα είναι ικανοί να διαχειριστούν δισεκατομμύρια ευρώ που θα έχουν στη διάθεσή τους για την περίοδο 2014-2020. Αυτά που είπατε όμως είναι σημαντικά. Είναι ζωτική η καινοτομία για πολλές περιφέρειες. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή τη στρατηγική εφιούς εξειδίκευσης, η οποία συμβαδίζει με τα ισχυρά στοιχεία μιας περιφέρειας. Σίγουρα το Smart Specialization δεν σημαίνει ότι όλες οι περιφέρειες μπορούν ε, να γίνουν Silicon Valley. Θα πρέπει όμως ε, να ε, βοηθήσουμε τις περιοχές αυτές στα ισχυρά του σημεία, είτε στον τομέα της υγείας, είτε στον τομέα ε, της ευρωπηγικής, στην Πολωνία ή στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων. Στην Ισπανία έχω επισκεφτεί πολλές ε, περιοχές και είδα παραδείγματος χάρη ότι αυτή η έννοια της ε, φιούς εξειδίκευσης μπορεί να οδηγήσει στο να συνεργαστούν ε, οι ακαδημαϊκοί με τη δημόσια διοίκηση και με τους ε, επιχειρηματίες προκειμένου να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη των περιφερειών. Για την ε, μεταναστευτική κρίση. Να σας πω το εξής. Εγώ ενεπλάκην από την αρχή. Καταρχήν συνεργάστηκα με τους δημάρχους έτσι ώστε καταρχήν τα κράτη-μέλη οι τοπικές αρχές ε, στα κράτη-μέλη είναι οι πρώτες που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Παρακολούθησα τη δραστηριότητα πολλών τοπικών αρχών που παραδειγματικά κινητοποιήθηκαν όταν έπρεπε να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό ζήτημα. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε και με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο ο οποίος μέσω του Ταμείου ΑΜΙΦ για το άσυλο και τη μεθανάστευση και την ένταξη ε, παρουσιάζει κάποια έκτακτα μέτρα και έχουμε και τη συμμετοχή του Κοινωνικού Ταμείου αλλά και του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια Ευρώπη ισχυρή που να τους συμπεριλαμβάνει όλους, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον ε, τα γκέτο, την ριζοσπαστικοποίηση των πολιτών μας κτλ. Έτσι λοιπόν τα ταμεία μας αποτελούν ε, έναν εξαιρετικό τρόπο για να συμβάλλουμε στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Στο Βερολίνο, παραδείγματο χάρη, επισκέφθηκα ένα, ε, τόπο ε, όπου έχουμε ένταξη των μεταναστών και αυτό γίνεται με ευρωπαϊκά κονδύλια και στο Άμστερνταμ έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο δημάρχων, ο δήμαρχος του Άμστερνταμ υλοποίησε αυτή την ε, εταιρική σχέση, όμως ε, δυστυχώς ε, κατέληξε και λυπάμαι γι' αυτό, πάθαινα και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί ουσιαστικά σύστησε αυτό το δίκτυο Τώρα ο Δήμαρχος της Αθήνας είναι επικεφαλής αυτής της εταιρικής σχέσης. Θέλουμε λοιπόν να καταλευτούμε όλες τις συνεργίες ε, μεταξύ των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεισφέρουν ε, και στη δημιουργία τοπικών συνεργειών. Το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ήδη έχει χρηματοδοτήσει κάποιους σημαντικούς τομείς, όπως η πρόσβαση ε, στην εκπαίδευση, στην έγκαιρη ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, ε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, κατασκευάσουν κάποιες κατοικίες αυτόνομες. Παρ' χάρη στο Μόλενμπεκ θαύμασε ένα σχέδιο, ένα project. Ξέρετε ότι οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τα κονδύλια από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, και τα έδωσαν στους γιατρούς χωρίς σύνορα που ασχολούνται με την ένταξη των μεταναστών στο Μόλενμπεκ ε, για να δημιουργηθούν δύο κέντρα στο Μόλενμπεκ, ένα στο Μόλενμπεκ και ένα στο Άντερλακτ. Αυτό συνέβη στην Ιταλία με την αλλαγή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Είχαμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ασφάλεια. Είδατε φέτος το καλοκαίρι δύο σκάφη που έσωσαν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στη Μεσόγειο. Αυτά αγοράστηκαν με ευρωπαϊκά χρήματα, τα σκάφη, αυτά τα πλοία. Οι Ιταλικές αρχές ε, αποφάσισαν ε, να ε, τροποποιήσουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την άμυνα και με ευρωπαϊκά χρήματα απέκτησαν αυτά τα σκάφη. Είμαστε πολύ ευέλικτοι λοιπόν. Είμαστε ανοιχτοί να αλλάξουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα. Το είπαμε στα κρατημέλη γιατί ξέρουμε ότι αυτή η πρόκληση δεν υπήρχε όταν έκλεισαν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Με την οθέτηση του Omnibus είμαι πεπισμένη ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο τα ευρωπαϊκά ταμεία για τέτοια ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη να μην διστάσουν να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε μια εταιρική σχέση σε σχέση με την ένταξη των μεταναστών. Ελσίνκι, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Βαρκελόνη, Αθήνα συμμετέχουν. Και έχουμε και μια λυσίδα Δανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία μια λυσίδα κρατών ε, και εμπειρογνωμονών από ΜΚΟ, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και έχουμε και μία άλλη πρωτοβουλία των αναπτυξιακών ταμείων. Περιμένουμε την ε, πρόσκληση υποβολής προτάσεων και την κατάθεση σχεδίων για να δούμε πώς γίνεται η ανταλλαγή των πρακτικών. Γιατί κάποια κρατημέλη έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε ό,τι αφορά την αντίξη των μεταναστών αναφέρομαι εδώ στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, ενώ άλλα κράτη πραγματικά έχουν κατακλειστεί και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εγώ έχω ε, επισκεφθεί κάποια νησιά, παραδείγματο χάρη ένα πολύ μικρό νησί που βρίσκεται στα 5 χιλιόμετρα απόσταση από την Τουρκία, με 5.000 κατοίκους και 9.000 μετανάστες με το δήμαρχο στη μέση, ε, και υπήρχαν απειλέ ε, τη μια μέρα από τους εντόπιου, την άλλη μέρα απειλές από τους μετανάστες. Καταλαβαίνετε την κατάσταση. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τι τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν τέτοιε καταστάσεις. Σε σχέση τώρα με τη συνεργασία μας με την ΟΛΑΦ. Να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε μία πολύ στενή συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης ΓΔΡΙΤΖΙΟ και της ΟΛΑΦ Έχουμε μια στρατηγική κατά της απάτης που έχει υπογράψει ο Γενικός Μα Διευθυντής για την περίοδο 2000 2015 2017 που καλύπτει 7 ευρωπαϊκά ταμεία και την πολιτική συνοχής. Έχουμε συχνές συναντήσει και πιστεύω ότι αυτή η καλή επικοινωνία έχει οδηγήσει στην αποσαφήνιση πολλών περιπτώσεων σε ό,τι αφορά τις παρατυπίε και είδαμε τι εντάσσεται στην απάτη ή τι εντάσσεται στην παραγνώριση των κανόνων. Όταν προσφεύγει σε μας η Όλαφ για κάποια υπόθεση, εμείς αμέσως ε, παρακολουθούμε την κατάσταση και αναστέλουμε τις πληρωμές και ξεκινάμε διαδικασίες ε, χρηματοοικονομικών διορθώσεων για να ανακτήσουμε κάθε ευρώ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2007-2013, όλες οι έρευνες της Όλαφ θα ε, δημοσιευτούν ε, και ε, στο τέλος της περίοδου, στο κλείσιμο της περίοδου, έτσι ώστε να προστατεύεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός από πιθανές απάτες ή παρατυπίες. Μου λέει ο κ. Φερέγκο ότι ξέχασα να σας πω, Πρόεδρε, για τα λάθη που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Να επανέλθω, γιατί μου είπαν ότι δεν έδωσε ολοκληρωμένη απάντηση στην ερώτησή σας για τα λάθη που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Να σας διαβεβαιώσω, Πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν είμαστε πάντοτε ικανοποιημένοι. Γιατί φυσικά πρέπει να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Όμως παρακολουθούμε ότι λειτουργούν καλά όλα τα συστήματα, αλλά φυσικά πρέπει να βασιζόμαστε και στα διάθεσιμα αποτελέσματα του ελέγχου. Όπως σας είπα, έχουμε 500 εκθέσεις ετησίως από τους εθνικούς ε, ελεγκτές και δεν έχουμε την ε, ικανότητα να κάνουμε όλους τους ελέγχους, αλλά στοχεύουμε σε όλα τα προγράμματα υψηλού κινδύνου για να δούμε ότι έχουμε υψηλή ποιότητα ελέγχου. Προσπαθούμε να οθήσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν ε, ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς και ξέρετε ότι διακόπτουμε αμέσως ή αναστέλουμε τις πληρωμές μόλις βλέπουμε σοβαρές παρατυπίες. Επίσης, έχουμε σχέδια δράσης για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να οικοδομήσουν εύρωστα συστήματα επαλήθευσης και να διορθώνουν τα προβλήματα. Σας διαβεβαιώ ότι αν δεν διορθωθούν οι δαπάνες και αν δεν διορθωθούν τα συστήματα δεν καταβάλουμε τις πληρωμές. Ξέρετε πολύ καλά ότι προσφέρουμε στοχευμένη υποστήριξη στις αρχές και έχουμε μία πρωτοβουλία ε, για την ε, ε, βελτίωση των ελέγχων, έχουμε κάποια εργαλεία βελτίωσης των ελέγχων, ε, κατάρτιση κτλ. Υπάρχουν κάποια λάθη που θα μπορούσαν ε, να έχουν αποφευχθεί στις δημόσιες συμβάσεις. Ε, σας είπα ότι το 70% θα μπορούσε να έχει ανιχνευθεί, γιατί αυτό αφορά την επιλεξιμότητα στο επίπεδο των διαχειριστικών ερχών θα μπορούσε να έχει ανιχνευθεί. Και να εργαστούμε σκληρά για να εφαρμόσουμε όσο θετήσαμε το 2017 σε σχέση με τις κριτικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την πλειονότητα των λαθών. Αυτή είναι τώρα μια κοινή απάντηση σε εσά Πρόεδρε και στην κυρία Νταμπάλοβα. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε πολύ αυστηρά την εφιστάμενη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό που βλέπω για δεύτερο, έτος, για δεύτερο συναπτό έτος ε, Τώρα ε, είναι η κύρια πηγή της των λαθών είναι η επιλεξιμότητα. Εξακολουθεί να παραμένει το θέμα των δημόσιων συμβάσεων η κυρία πηγή σφαλμάτων σε κάποια κράτη-μέλη. Και πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Κύριος Τσεχόφσκι. Καλά το από το όνομά σας. Θα ήθελα να σας ε, δώσω μια μονολεκτική αρνητική απάντηση. Έχουμε την ίδια προσέγγιση ε, ως προς ελέγχους στα κράτη-μέλη, όχι διαφορετικούς, με τον κανονισμό, με τη μία διαδικασία. Ε, μετά μιλήσατε για το gold plating, για την προσαρμογή στις ε, προτιμήσεις των κρατών μελών. της οδηγίας που συνοδεύτηκε από χιλιάδες σελίδων ε, με την ένδειξη ότι αυτό ζητούσαν οι Βρυξέλλες. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς δεν ζητούμε 100 ε, ή 500 σελίδες ε, για ένα project και στο χώρο των σιδηροδρόμων έχουμε δει και project με 10.000 σελίδες υπογεγραμμένες μία-μία ή μονογραμμένες μία-μία. Δηλαδή αντί για εφαρμογή βάζουν υπογραφές. Πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν με τις ε, χώρες. Ικανότητα απορρόφησης επίσης. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει απλοποίηση. Μίλησα για το την επιλογή απλουστευμένου κόστος, τα χρηματοοικονομικά μέσα και την ε, εισαγωγή σε αυτό που λέμε πολιτική συνοχής. Πιστεύω ότι ως ε, συνέπεια των συστάσεων της ομάδας για την περίοδο μετά το 2020 μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή των ε, δικαιούχων. Όμως, χωρίς τις προσπάθειες των κρατών μελών, δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα το καταρθώσουμε. Γιατί όταν ε, μιλάμε για απορρόφηση και για εφαρμογή, την ευθύνη την έχουν 100% ε, τα κράτη-μέλη. Ούτε εσείς από το Κοινοβούλιο, ούτε εμείς από την Κομισιόν δεν μπορούμε να πάμε επί τόπου και να υλοποιήσουμε την εφαρμογή των σχεδίων. Πιστεύω ότι είναι φιλοδοξία του, του κάθε κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι φιλοδοξία του κάθε κράτους μέλους, να υποφεληθεί από αυτή την ε, μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη της χώρας του. Πρόκειται για μια ευκαιρία που θα μπορούσε να είναι και η τελευταία στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αν θα μπορούν να αποφελουθούν και στο μέλλον τα κράτη-μέλη. Εμεί θέλουμε να έχουν περισσότερα κονδύλια τα μέλη από τα διαφορετικά ταμεία, αλλά θα πρέπει και αυτά να συνειδητοποιήσουν ότι αν δεν μπορέσουν ε, να δείξουν στα χαρτιά ότι είναι σε θέση να δαπανίσουν αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται ως μια χειρονομία αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, θα μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγωνιστούμε για μια πολιτική συνοχής στο επίπεδο που την έχουμε και σήμερα. Κύριο Βόγκαν. Νομίζω ότι έθεσε ένα πολιτικό πρόβλημα, πολύ σοβαρό. Η πολιτική συνοχή είναι πολιτική δαπανών που επενδύει δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό δικαιούχων που είδαν σε αυτή την πολιτική μια ευκαιρία ε, απάτης. Και μέσω των υποθέσεων που δημοσιεύτηκαν και αναδημοσιεύτηκαν τροφοδοτήθηκαν ε, κάποιες υποψίες ε, για το σύνολο της ε, πολιτικής. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μόνο 0,7% των πληρωμών της πολιτικής συλλογής για την περίοδο 2007-2013 σε ό,τι αφορά τις απάτες. Έχει μηδενική ανοχή η Κομισιόν απέναντι στη διαφθορά και στην απάτη και κάθε φορά που ανοιχνεύουμε κάποιες περιπτώσεις έχουμε υποψίες, λαμβάνουμε μέτρα. Άκουσα τι είπε ο κ. Βόγκαν, δεν σημαίνει ότι τα λάθη, τα σφάλματα είναι και απάτη. Όταν μιλάμε για παρατυπίες μπορεί να έχουμε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενώ η απάτη είναι κάτι σκόπιμο η οποία υποσκάπτει τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, Όλαφ, γιατί ήταν εδώ την προηγούμενη Δευτέρα και μας είπαν ότι 90% των απατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίζονται στα διαφορετικά ταμεία. Άρα χρειάζεται πιστή προσοχή αυτή η υπόθεση. Και ένα ουγγρικό πρόγραμμα ήταν νομίζω. Εκείνο που παρουσιάστηκε σαν ε, παράδειγμα. Για να δούμε αν μπορούμε να αναζητήσουμε τα κονδύλια. Κυρία Ιβάνοβα έχει το λόγο παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη θέση μου. Ωστόσο, ε, ε Ήγηραν πολύ ενδιαφέροντα θέματα οι βουλευτέ σα. Ξεκινήσω με τον κύριο Τσέλερ που αναφέρθηκε στη σημασία τη συνοχή για την προαγωγή τη ανάπτυξη και, της θέσης, και των θέσεων απασχόληση το ποσοστό σφάλματος και καθυστερήσει στην νέα προγραμματική περίοδο με βρίσκουν σύμφωνοι και τα ζητήματα σχετικά με την απορρόφηση. Εδώ θα ήθελα κύριε Τσέλερ να σας ενημερώσω ότι θα υπάρξει ειδικό τμήμα ε, στην έκθεση από το δεύτερο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα δημοσιευθεί το προσεχές έτος, ειδικά για το θέμα της απορρόφησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους λόγους των καθυστερήσεων και προτάσεις για αντιμετώπιση τους. Επί τη ευκαιρία λοιπόν σας κάνω και τη διαφήμιση της έκθεσής μας για το σημαντικό αυτό θέμα επίσης. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τις ε, διαδικασίες των ε, προμηθειών, των ελέγχων, συγγνώμη, εδώ έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα προφανή ζητήματα. Ο έλεγχος δημοσιονομικός ήδη βλέπουμε να πολλαπλασιάζεται και υπάρχουν ακόμη και ε, μελέτες σε πανεπιστημιακό επίπεδο που χρησιμοποιούν τον όρο έκρηξη δημοσιονομικού ελέγχου πλέον, εκρηκτικές δεστάσεις δηλαδή έχουν λάβει. ως εξωτερικός δημοσιονομικής ελεγκτής εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στην ε, σειρά ή στην αλυσίδα τον κύκλο των εσωτερικών δημοσιονομικών λεκτών όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο θα προσπαθήσουμε με ένα πλειοτικό πρόγραμμα το προσεχές έτος να επαληθεύσουμε εάν μπορούμε σε συγκεκριμένο χώρο στη συνοχή να επαληθεύσουμε τη δουλειά που κάνουν άλλοι και να δούμε αν είναι δυνατόν να εξετάσουμε και την, ε, να αποκαταστήσουμε και το υπολοιπόμενο ποσοστό λάθους σε σχέση με την δήλωση συμμόρφωσης. Επίσης, τα δημοσιονομικά οι πράξει μουσονομικέ, οι άμεσε έχουν ασφαλώ πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, αλλά θα σα υπενθυμίσω ότι είναι υπαριθμόν 19 ειδική έκθεση του 2015 για, τα, για τις δημοσιονομικές πράξεις ε, για τα δημοσιονομικά νομοθετήματα που έχουν προβλήματα ε, και όγκου, καθυστέρηση στην εφαρμογή, ε, κόστους, αλλά βέβαια και λογοδοσίας για την οποία διατυπώνουμε συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πληρέστερες πληροφορίες για το κόστος και τα τέλη για τη, της διαχείρισης, διεξαγωγής συγκριτικής ανάλυσης στο κόστος των ε, δανείων και των άλλων δημοσιονομικών μέσων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και των νομοθετημάτων που θα μπορούσαν να προετοιμαστούν για την περίοδο του μετά το 2019. με την προσφορά και τεχνογνωσία τη τεχνικής υποστήριξη. Στην ερώτηση κυρία Λαπάγιοβα, και αλλά και τη δική σα για τι δημόσιε προμήθειες μπορώ να πω ότι ω ελεγκτική αρχή ελέγχουμε εκ των υστέρων γεγονότα, έργα, σχέδια εάν ε, επιτελούν τον, ε, τον ε, δεδηλωμένο στόχο τους. Από εκεί πέρα είναι πολιτική επιλογή αν θέλετε εκ των προτέρων επαλήθευση. είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει σε δύο ειδικέ εκθέσεις, αλλά δεν ε, καλύπτεται από τις γενικές μας εκθέσεις επαληθεύσης επίσης, της δράσης της διαχείρισης που άλλωστε και η Επιτροπή επισημαίνει ως προς την ανεπαρκή κάλυψη των επαληθεύσεων από τη διαχείριση της δράσεως των ε, ενδιαμέσων ε, διαμεσολαβητών. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του διαγνώσιμου λάθους. Δαπάνες του 2013 μπορούν να δηλωθούν τελευταία φορά φέτος και ως εκ τούτου μία δραστηριότητα που έχει υποβληθεί σε επαλήθευση της δράσης της διαχείρισης μπορεί να εμφανίζεται πιο συχνά στο, στις εκθέσεις μας. Αυτά σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, για τις εκθέσεις μας, για, ε, για, για τις μας. Ευχαριστώ και για να κλείσουμε πάρα πολύ στο μάο κύριο Τσέλερ. Πρόεδρε... Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η πολιτική των, των διαρθωτικών αλλαγών ε, και η πολιτική συνοχή ε, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρέπει να δούμε τώρα τις προγραμματικές περιόδους και διαπιστώνουμε ότι εντωμεταξύ για τα κράτη-μέλη αλλά και για τις ε, οι αλλά και άλλες εταιρείε έχουν ε, διαφορετικές δυνατότητες ε, χρηματοδότησης που είναι πιο ελαφρές διοικητικά από τα διαφορετικά ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μιλά για 60 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε δάνεια, μάλλον μηνιαίως 60 δις δάνεια και ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Οδηγικές Επενδύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων είναι στη διάθεση να κρατών μελών. Οπότε, ε, μάλλον ε, παίρνει δεύτερη θέση το, η χρήση των διευθυντικών ταμείων. Βεβαίως, όταν μιλούμε για τις δημοσιονομικές αρχές και την διόρθωση, εξέταση των λαθών, αυτό θα μπορούσε να είναι ε, ενδιαφέρον για να μπορούμε να αποκλείσουμε την αρχή τα λάθη τα οποία θα οδηγούσαν σε επιστροφή ήδη ε, καταβληθέντων ποσών. Αλλά βεβαίως η έκθεση λέει ότι όταν βάζουμε κάποιους συμβούλους εταιριών σε αυτούς τους ελέγχους, ε, εξετάζουν πραγματικά πολύ αυστηρά το πώς γίνονται η συμπλήρωση και πώς διορθώνονται τα λάθη. Δείχνουν δηλαδή ότι παίρνουν σοβαρά το ρόλο τους. Έτσι ώστε να μην ε, υπάρχει ε, δυνατότητα να ε, ξαναέρθουμε σε διαδικασία παρέμβασης από το Ταμείο. Τώρα, για το 2018 και τα περαιτέρω κονδύλια, να σας πω ότι το 2015 είχαμε 70 ε, δισεκατομμύρια τα οποία ήρθαν πίσω στον Ευρωπαϊκό Κοργανά. Τώρα έχουμε ένα αντίστοιχο ποσό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Στο Στρασβούργο, με την επίγουσα διαδικασία, αποφασίσαμε μια, μια διαφοροποίηση των ε, διαδικασιών για τα διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, να μπουν δηλαδή εκεί τα κονδύλια. η οποία δουλεύει αρκετά αποτελεσματικά και εντατικά. Αυτό όμως που με ενοχλεί κάπως είναι βεβαίως ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, ορατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τι κάνουμε με τα μέσα αυτά τα οποία μέχρι στιγμής δεν, τα οποία μπορεί να μην είναι σε διαθέσιμα στο επίπεδο που ήταν μέχρι τώρα. Θα πρέπει να τα καταστήσουμε πιο διαθέσιμα και να επιταχύνουμε τη διαδικασία και στις περιφέρειες. Διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλές καλές πρωτοβουλίες, προσεγγίσεις ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την έρευνα, και εκεί μπορεί να υπάρξει πρόοδος, κυρίως ό,τι φορά το πλεόνασμα από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς όμως στο διοικητικό επίπεδο υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Όπως είπαμε σήμερα αρκετές φορές και δυστυχώς τα κονδύλια δεν φτάνουν εκεί που πρέπει. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε για να βελτιώσουμε, διότι πραγματικά το τέλος της προγραμματικής περίοδου βρίσκεται πάρα πολύ κοντά μας. Βεβαίως θα παραμείνουμε σε επαφή με την Επίτροπο. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας εδώ, για τις προφορικές σας απαντήσεις, για τις γραπτές σας απαντήσεις. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό και βεβαίως σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και τώρα να καλέσουμε τον ε, πρόεδρο του ε, ελεγκτικού συνεδρίου να του ζητήσουμε και ένα συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε. να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων για το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Ελεκτικού Συνεδρίου. Παρακαλώ, συνάδελφοι αν μπορείτε όχι τόσο θόρυβο, παρακαλώ αποχωρήστε ησύχω για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είστε εδώ για να συζητήσουμε για το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι εντυπωσιακό το πρόγραμμα εργασίας σας. Ε, είδαμε την ειδική έκθεση. Έχουμε 12 ειδικέ εκθέσεις οι οποίε εντάσσονται στην, ε, στην ε, έκθεση του προηγούμενου έτους. Βλέπετε εδώ με κόκκινο. Βεβαίω τώρα το ερώτημα είναι πόσο αξιόπιστο είναι το πρόγραμμα εργασία ε, του ελεγκτικού συνεδρίου με τι εκθέσει εκθέσεις οι οποίε έρχονται γέρο με αυτέ που δεν έρχονται γέρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Καταρχά, να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα στην αρχή. Το πρόγραμμα εργασία είναι ένα πρόγραμμα εν εξελίξη. Ένα έργο εν εξελίξη. Οι δηλαδή που κάνουμε, καμιά φορά όταν προετοιμάζονται ή όταν ολοκληρώνονται, αντιμετωπίζουν ε, κάποια απρόπτα. Κάποιες απρόπτε συνθήκες, ε, οι οποίες οδηγούν σε καθυστερήσεις γιατί δεν είναι τα διαθέσιμα τα έγγραφα εγκαίρω, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την αρχή. Προσπαθούμε φυσικά πάντα να το αποφύγουμε αυτό, να βελτιώσουμε τις συνθήκες και στα σεμινάρια και που έχουμε οργανώσει και το Σεπτέμβριο φέτος υπήρξε το ερώτημα αυτό της επεξεργασίας της μεθοδολογίας για το πώς διαχειριζόμαστε όλες αυτές τις εκθέσεις και επίσης η Επιτροπή Ποιότητας των Εκθέσεων θα δούνε όλα τα εγχειρίδια, όλες τις λεπτομέρειες για το πώς μπορούμε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα να διεκπεραιώνουμε τις έκθεσεις έτσι ώστε εγκαίρως να είναι στη διάθεσή μας. Ποτέ δεν χάνεται μια έκθεση. Κάποια στιγμή όμως φτάνει στο τραπέζι μας για συζήτηση. βέβαια, θα προσπαθήσουμε εμείς να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και το χρονοδιάγραμμα να το τηρούμε. Για το πρόγραμμα εργασίας 2018. Τον Οκτώβριο το δημοσιεύσαμε. 15 project έχουμε περίπου, τα οποία αναφέρονται εδώ στο πρόγραμμα εργασία. Υπάρχουν βεβαίω ε, πολλέ ε, δημοσιεύσει, ειδικέ εκθέσει, αιτήσει εκθέσει, θεματικά ε, έγγραφα, γνωμοδοτήσει. Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα λοιπόν βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ανάπτυξη και ένταξη, μετανάστευση και παγκόσμια ανάπτυξη, εσωτερική αγορά και Ευρωπαϊκή Ένωση της Οικονομίας και της Λογοδοσίας. Για το 2018 έχουμε και κάποιες νέες πρωτοβουλίες, έχουμε υψηλής προτεραιότητας πρωτοβουλίες και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να τις ε, ε, δημοσιεύσουμε στο ε, πρόγραμμα για το 2018. Ας πούμε, το μέλλον για την κοινή αγροτική πολιτική, η απλούστευση της, κοινωνικής, της πολιτικής συνοχής, η απλούστευση του ορίζοντα 2020, ε, ασφάλεια τροφίμων επίσης, ε, διαφάνεια της ε, χρηματοδότησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάτι που το ζήτησε η Επιτροπή σας έντονα, διευκόλυνση για τους πρόσφυγες από την Τουρκία, μια έκθεση για, την, για τη δεοντολογία και, και την επίλυση διαφορών. Επίσης, με βάση και τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ένωση, και τους ε, κινδύνους που λαμβάνουμε, ένα σημαντικό κριτήριο για, την, για τον καθορισμό των εκθέσεων είναι και οι δικές σας απόψεις ε, που έχουν να κάνουν φυσικά με, την, ε, με τις απαλλαγές. Έχουμε την, τον κατάλογο για τις διασκέψεις. Από τον κατάλογο τώρα των διασκέψεων αυτών για το 2018 έχουμε περίπου 2 τρίτα των προτάσεων τα οποία έχουν, καλύπτονται είτε με ήδη ολοκληρωμένες εκθέσεις, είτε με εκθέσεις που βρίσκονται να εξελίξει. Οι προτάσεις οι περισσότερες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή σας και βρίσκονται στον κατάλογο αυτών των διασκέψεων. Έχουμε στείλει μια επιστολή στην Επιτροπή Βίξτρομ με όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα, για τις επιθυμίες που υπάρχουν, για το πρόγραμμα το περσινό, έλειπε η συμβολή κάποιων μεγάλων επιτροπών ή, εν πάση ήρθε πάρα πολύ αργά. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσετε αυτές τις ε, επιτροπές να τους, ε, να τους επιστήσουμε την προσοχή στο πόσο σημαντικό είναι εγκαίρως να υποβάλουν τις προτάσεις τους για να μπορούν να καταλήγουν αυτές σε συγκεκριμένες εκθέσεις. Μετά, για το πρόγραμμα εργασίας, προετοιμασία. Έχει ήδη ξεκινήσει. Η επόμενη συνάντηση είναι η διάσκεψη των Προέδρων για τις 16 Ιανουαρίου του 2018. Σίγουρα εκεί θα δούμε τις πρώτες ιδέες για το πρόγραμμα εργασίας 2019 ήδη. Αυτά συνοπτικά. Το πρόγραμμα εργασίας μας ε, πρέπει να το έχετε λάβει και γραπτός. Να σας ευχαριστήσω, για, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας μάλλον για την πολύ εντατική και πολύ καλή συνεργασία που έχουμε για την προετοιμασία, για τη διεκπαιρέωση, για την εφαρμογή. Ξέρω ότι βεβαίως ε, και από τη δική μας την πλευρά πάντα υπάρχουν σημεία που υπάρχει δυνατότητα βελτίωση. Το είπα και την προηγούμενη ε, εβδομάδα στην ε, διάσκεψη των Προέδρων, αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τα που θα προσπαθούμε να τα λύσουμε, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε εν μια ανοιχτή μπορεί να ολοκληρωθεί. Αυτά προς το παρόν ήθελα να σας πω. Αν υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις, ευχαριστώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για την πολύ καλή συνεργασία. Πάντοτε εισακούονται οι επιθυμίες μας στο πρόγραμμα εργασίας. Είναι τεράστια η ευκαιρία που έχουμε να δούμε και την υλοποίηση στο τέλος του χρόνου των προτάσεων μας σε σχέση με τις εκθέσεις αναχώρα. Θέλω να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικές, διότι και στις διάφορες ε, επισκέψεις μας βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι, όπως άλλωστε και σήμερα, και με το ερωτηματολόγιο προς την ε, Επίτροπο, αλλά και το ερωτηματολόγιο που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε πλειοδοσίες από έναν μόνο πλειοδοτούντα ε, σε κράτη, πολλές σε πολλά κράτη. και μάλιστα από το κράτο το ίδιο, άρα δεν έχει ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Άρα είναι πολύ σημαντικά τα θέματα, δεν μπορούμε να τα παραμελήσουμε και επανέρχομαι με αυτό, χωρίς να έχω πρόθεση να καταγγείλω, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και θέτει αμφιβόλω τελικά και την εξυπηρέτηση των στόχων και την ίση μεταχείριση. Νομίζω ότι οι εκθέσεις αναχώρα μπορούν να δώσουν μια πραγματική εικόνα των προβλημάτων ε, στις πραγματικές τους διαστάσεις και αντίστοιχα αναλόγως των διαστάσεων να δοθεί και κατάλληλη λύση. Και βέβαια με πάντα εκκρεμές το ερώτημα πώς θα δημορφωθεί ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το κεφάλαιο ειδικά της γεωργικής πολιτικής. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν ορισμένοι, ενώ ο κόσμος ολόκληρος αλλάζει, να λένε ότι δεν μπορεί να αλλάξει καν ε, η γεωργική πολιτική. Ο κύριος Λένε, σε σχέση με, την, με τις εκθέσεις χώρα, προσπαθούμε όντως να τις βελτιώνουμε κάθε φορά. Ξέρετε, ότι είχαμε στο παρελθόν προβλήματα σε σχέση με τις στατιστικές πληροφορίες ε, που ήταν διαθέσιμες για τις εκθέσεις μας κατά τη διάρκεια του έτους. Ήταν δύσκολο δηλαδή να εκδώσουμε αξιόπιστες εκθέσεις ανά χώρα. Πάντως πιστεύουμε ότι με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα καταρτίζεται από εδώ και μπρος η έκθεση θα έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε και πρόσθετες πληροφορίες έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και των κατά χώρα αναχώρα εκθέσεων και με το performance reporting νομίζω ότι θα μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις ομαδοποιημένες χώρες αλλά και για επιμέρους χώρες. Στο συγκεκριμένο όμως θα έχουμε ομαδοποιη... ομάδες χωρών, χωρίς δυσκολία μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Με το performance reporting θα διαπιστώσετε ότι και στο παρελθόν το έχουμε κάνει, δηλαδή έχουμε δώσει έμφαση σε ένα συγκεκριμένο τομέα και έτσι σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουμε ε, ενσκήψει και έχουμε εξετάσει συγκεκριμένα τι προβλήματα μπορούν να υπήρχαν. Επίση, στη διάσκεψη των ε, Προέδρων, είπα την προηγούμενη εβδομάδα και το παραλαμβάνω και εδώ, ότι θα υπάρξει ένα ε, πρώτο έγγραφο ενημέρωση στα τέλη Ιανουαρίου, το πολύ αρχά Φεβρουαρίου, στη διάθεσή σα και άπαξ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύσει τι προτάσει τη σχετικά σύντομα, μέχρι το καλοκαίρι, θα έχουμε τοποθέτηση για το πολιτές οικονομικο πλαίσιο με τη γνωμοδότησή μας, η οποία ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη. Οι τάσεις ε, που θα επιλέγουν ε, δεν ε, είναι δυνατόν να εκτεθούν αυτή τη στιγμή, αλλά αν έχετε δει τα προηγούμενα μας έγγραφα, θα έχετε αντιληφθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στη διαφάνεια, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και οπωσδήποτε και το τομέα τη Γεωργία θα βρει τη θέση του σε αυτέ τι προτάσει. Για το πρόγραμμα εργασία του δικό μα ε, του επόμενου έτου ήδη προβλέπουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα τη της ε, Γεωργία ε, στι εκθέσει μα και ιδιαίτερα σε σχέση με τις μεγάλες προκλήσεις σχετικές με τη γεωργική πολιτική στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, των οποίων έχουμε πλήρη συνείδηση και επ' αυτού βέβαια αναπτύσσονται και οι συζητήσεις στο ελεγκτικό συνέδριο και πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε με τη δική μας συμβολή στη βελτίωση της συζήτησης και την επιτάχυνση των εργασιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τώρα εγώ θα εκπροσωπήσω μάλλον την Πρόεδρο. Κυρία Γεράσεντερ, έχει το λόγο για τις ερωτήσεις της. Δεν ε, κοιτούσα το Προεδρείο και ξαφνικά είδα ξαναμίστη, κυρία, κυρία Γκρέσλε. Βέβαια θα μου άρεσε να την είχα ακούσει γιατί αυτή λέει ότι είμαστε ε, σε αυτή την επιτροπή ε, όλοι ε, τρελή να ακούμε πώς ε, ασκούμε κριτική σε κάποιες χώρες. Ότι μας αρέσει πολύ να ασκούμε κριτική. Όμως ε, δεν βρισκόμαστε όλοι σε αυτή τη θέση και μάλιστα τα 8 μέλη της δικής μου επιτροπής. Ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις ιστορικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Βορράς και Νότου και Ανατολής και Δύσης. Να μην ε, κάνουμε τέτοιες ε, κριτικές. Εγώ βέβαια γνωρίζω ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει πολύ μεγάλη ικανότητα ε, να παρουσιάζει με ιδιαίτερα ουδέτερο τρόπο τις πολιτικές του αναλύσεις σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επομένως, Θα ήθελα να μην κάνουμε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ καλών και κακών με τέτοιο απλουστευτικό και λανθασμένο τρόπο. Γιατί αντί να βοηθάμε τελικά ε, δεν συνεισφέρουμε. Αντί να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε λύσεις, αν ε, παίρνοντα χάρη βλέπαμε κάποιον υπουργό και κάναμε διάλογο, τότε ήταν επικοδομητικό. Ενώ αν ε, πάντοτε κατηγορούσαμε τους ανθρώπους για τα ίδια, σταμάτησαν να έρχονται οι υπουργοί και χάσαμε σημαντικούς συνομιλητές. Στο πρόγραμμα εργασίας σας και στον τρόπο που λειτουργείτε, και στο γόητρο που δίνετε στο θεσμικό σας όργανο, νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ξέρω ότι οι ελεγκτές θέλουν να κάνουν τον κλασικό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτό το προϊόν ε, που εσείς ε, ε, ουσιαστικά το χρησιμοποιείτε για να γίνει μία αναθεώρηση, μία επισκόπηση όλων των δράσεων του ελεκτικού συνεδρίου συνέχεια είναι πολύ σημαντικό ε, να δούμε εμείς που έχει γίνει πρόοδος, που δεν έχει γίνει πρόοδος, που είναι τα θετικά σημεία που πρέπει να συνεχίσουμε να οθούμε και να μην ε, ξεχνάμε και σημαντικά προβλήματα που ανέκυψαν στην κοινή αγροτική πολιτική, στο Ταμείο Συνοχής ε, και σε άλλα σημαντικά ζητήματα. Και να δούμε πώς τα νέα θέματα, όπως η άμυνα, ή το μεταναστευτικό και προσφυγική κρίση και την αντιστάθμιση που αναζητούμε στην αναπτυξή συνεργασία, πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση των προσφύγων και των μεταναστών, χρησιμοποιώντας και άλλες πολιτικές Παραδείγματο χάρη είχαμε κάποιε ε, πολιτικές ε, στο θέμα της άμυνας, στην ε, πολιτική της επίλυσης των συγκρούσεων ή την πολιτική ίδρυσης περισσότερων πρεσβειών. Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όσα μας παρουσιάσετε για το 2018, δηλαδή όλο αυτό το θέμα της ε, δημιουργίας ε, θέσεων εργασίας, γιατί βλέπουμε ε, πολλές φορές ότι υπάρχουν ε, πολλά καλά παραδείγματα ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας και διατηρούνται και αυτές οι θέσεις εργασίας. Ή το θέμα του προϋπολογισμού που αφορά την ισότητα των δύο φύλων, το πώς εφαρμόζεται όπου βλέπουμε κάθε φορά ότι σε μία όλο και πιο γυρασμένη Ευρώπη ε, να πετύχουμε ε, το να πετύχουμε το είναι ένταξη 100% των γενικών στην αγορά εργασίας ε, ακόμη συναντά προβλήματα. Προλίγου συζητήσαμε και με την κυρία Κρέτσου. Αυτή η Επιτροπή προσπαθεί να δει πόση η δυναμική που έχει δημιουργηθεί με τα κράτη-μέλη και με την εμπλοκή τους ή όχι στην εφαρμογή των πολιτικών, με τις ακόλουθες συστάσεις, ουσιαστικά ε, γίνεται ε, ουσιαστικά ένα τεστ συνείδησης και όλα αυτά πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς θετικά. Πώς δηλαδή θα μπορούσαν αυτές οι συστάσεις ε, αναχώρα που κάνει η Κομισιόν και που υιοθετεί το Συμβούλιο, πώς ε, θα μπορούσαν να προωθηθούν και από το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί σε ορισμένες χώρες ε, μπορεί τελικά να υλοποιούν τα καθήκοντά τους, όμως τελικά βλέπουμε ότι το Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο μπορούν ε, να βοηθήσουν ε, τις χώρες που έχουν άλλες δυσκολίες να βελτιωθούν. Και ξέρετε τώρα σε ποιες χώρες ε, αναφέρομαι. Ίσως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιες από αυτές τις χώρες να μπλοκάρουν μία κατάσταση που δημιουργεί συνεχώς σε όλους εμάς προβλήματα. Δηλαδή κάποιες χώρες ε, έχουν ε, μόνιμο πλεόνασμα ε, και οι επενδύσεις στην παιδεία, στην υποδομή ουσιαστικά θα μπορούσαν να γίνουν και εκεί όπου λείπουν. Δηλαδή θα μπορούσαν οι χώρες αυτές να μας βοηθήσουν να λειτουργήσει καλύτερα και η υπόλοιπη Ευρώπη. Θα έλεγα λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συστάσεις που επαναλαμβάνονται στο εξάμεινο έτσι ώστε να μπορέσει το ηλεκτρικό συνέδριο να μας βοηθήσει και με τη δική του εμπειρία και με τα δικά του εργαλεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράνκα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ που παρουσιαστήκατε εδώ σήμερα ενώπιόν μας για να μας εξηγήσετε τις προτεραιότητες ε, του προγράμματος εργασίας για το 2018. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη κατά κάποιο τρόπο την ε, θεμελιώδη αποστολή του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγώ πιστεύω ότι ο κύριος στόχος είναι να προωθήσει την αποδόση να αυξήσει τη διαφάνεια και τελικά να δώσει τα στοιχεία έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους δαπανώνται σωστά. Το είπε και η κυρία Αγιάλα. Μόλις είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, για την απαλλαγή του 2016 με την Επίτροπο Κρέτσου έχει ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει πολύ σημαντικά ποσά, 35-36 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό, Πρόεδρε, να δούμε και την συλλογική εικόνα αυτών των δαπανών και να δούμε σε ποιες διαστάσεις κινούμαστε αφενός. Σε ό,τι αφορά τους ε, φυσικούς πόρους μιλάμε περίπου για 60 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίων στο γενικό πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην το χάσουμε αυτό από το νου μας. Ε, νομίζω ότι το ελεκτικό συνέδριο μπορεί να κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά σε ό,τι αφορά στο να παράσχει στις βουλές, ε, στα θεσμικά όργανα, σε σχέση με το πώς δαπανάται το σύνολο του προπολογισμού, ποιες είναι οι προτεραιότητες και σε ποιο βαθμό αντιμετωπίζονται κοινέ προκλήσει. Παραδείγματο χάρη στο θέμα τη ασφάλεια, το έφερε και η κυρία Γιάλα. Αν συγκρίνουμε τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέραμε, δηλαδή τι ε, πολιτικέ που αφορούν τα διεθνικά ταμεία ε, ή ε, τους φυσικούς πόρους, θα δούμε ότι υπάρχει μία πολύ μειωμένη τάση σε έναν τομέα που αφορά την ασφάλεια. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι τα έγγραφα του λεκτικού συνεδρίου θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να δώσουν νέο προσανατολισμό στις πολιτικές και για να μας θέσουν σε επαφή με την πραγματικότητα και με τα αιτήματα των πολιτών μας. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτα τα εγγραφά σα. Και ξέρω ότι έχετε και πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εργασία. Έχετε περίπου 900 άτομα που βοηθούν το ελεκτικό συνέδριο. Πώς λοιπόν θα αξιολογούσατε ε, το μέγεθος των προκλήσεων, τη φιλοδοξία των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν εδώ, σε σχέση με τους ανθρώπινους σπόρους που έχετε διαθέσιμους. Έχω και εδώ το πρόγραμμα έκθεσή σας, ε, συγγνώμη την, ε, το πρόγραμμα εργασίας σας για το περσινό έτος, πέρσι το ελεκτικό συνέδριο παρήγαγε 36 ειδικέ εκθέσεις Έχουμε και τις γνωμοδοτήσεις, τις συγκεκριμένες εκθέσεις ε, για τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πέρσι δημοσιεύσατε 52 εκθέσεις ε, και τις αναλυτικές δημοσιεύσεις, έγγραφα, πανοραμικές και φυσικά πέρα από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Πώς αυτό το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του 2018 τοποθετείται σε σχέση με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το οποίο μας ενημερώσατε πέρσι. Δηλαδή με ποσοτικού όρου, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο φιλόδοξο, γιατί είμαστε σε μια πιο ευαίσθητη στιγμή στο χρονοδιάγραμμα, αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών, ε, νέο κύκλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανθρώπινοι πόροι που εσείς διαθέτετε για αυτό το πρόγραμμα αρκούν ή δεν αρκούν. Προσαρμόζονται στο πρόγραμμα εργασίας σας. Εμένα με ενδιαφέρει ιδίω η εξωτερική εργασία σα. εμενα με ενδιαφερει Είμαι και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξωτερική πολιτική. Ποιες ε, προτεραιότητες δίνονται στην αξιολόγηση των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μιλώ μόνο για αποστολές παρατήρησης των εκλογών, αλλά και για αποστολές υποστήριξης, όπως το Σαχέλ, παραδείγματος χάρη. Πώς ε, βλέπετε, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά στο σύνολο των ε, δράσεων που παρουσιάσετε για το 2018. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Είμαι και εγώ στο κατάλογο των ε, ομιλητών. Έχω συγκεκριμένη σύντομη ερώτηση από τη Σκοπιά όμως περισσότερο των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε πολλά ακούσει για τις προτεραιότητες. Περιμένω βέβαια και τις απαντήσεις σας. Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη συνεργασία σας με τις τεχνικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις λοιπές κοινοβουλευτικές επιτροπές, γιατί μπορεί να σας εμπνέουν τα αιτήματα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αλλά οι τεχνικές σας ενδιαφέρουν. Έχετε επαφές συχνά με την Σεσίλια Βίξτρομ, την πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων και με τη Διάσκεψη των Προέδρων Πώς βλέπετε λοιπόν ε, το ενδιαφέρον των λοιπόν βουλευτών του Κοινοβουλίου για τη δουλειά σας. Α, και έχω και τον κύριο Σαρβάμα και θα σας δώσω το λόγο για τις απαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ. Λυπούμε που έχασα το πρώτο και μεγάλο μέρος της παρουσίασης σας, ε, κύριε Λένε. Αλλά από την άλλη θα πω ότι είναι τα ίδια, τα γνωστά αυτά που είπατε. Δεν βλέπετε και το καινούριο. Η έμφαση που εσείς έχετε δώσει από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου για τα επόμενα χρόνια ε, εστιάζεται στην αξιολόγηση των επιδόσεων και γι' αυτό σκόπιμο θα ήταν σήμερα να μας πείτε και το 2018 πιο συγκεκριμένα Τι προβλέπετε να μπορέσετε συγκεκριμένα να βελτιώσετε σε σχέση με το 17. έχω μια συγκεκριμένη περίπτωση υπόψη. Ε, είμαστε στη δικασία της απαλλαγής. Με ένα λοιπόν συγκεκριμένο παράδειγμα. με τα AMPRs, ε, τις διαχειριστικές αρχές. Και είχαμε και την Επίτροπο Κρέτσου εδώ. Ε, περισσότερο περιγραφική εικόνα βλέπουμε και όχι πραγματική αξιολόγηση και ξέρω ότι σας λέω τον ίδιο χαβά πάντα αλλά θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Λένα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Άγια Λαζάντερ αναφέρθηκε στο θέμα των ε, αναχώρα εκθέσεων και θέλω να καταστήσω σαφές εδώ. Προσπάθησα να το εξηγήσω ότι από τις στατιστικές που έχουμε στη θέση μας στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δεν είμαστε θέση να κάνουμε προβολές ανακράτος, αναχώρα, συγκεκριμένη συναλλητική και στατιστική μέθοδος που ακολουθούμε μας υποχρεώνει σε μια ε, συνολική έκθεση και όχι, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο κράτος. Δεν είναι εφικτό. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και διαρκώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε την κατάσταση είναι να συμπληρώνουμε ε, με ε, πληροφορίες αναχώρα συγκεκριμένες, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί ε, ενημέρωση, ανάλυση αναχώρα για το ποσοστό του σφάλματος. Απλώς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε προς τη διαφάνεια προς την μεθοδολογία που ακολουθούμε και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε νομίζω μπορέσει και με καλά αποτελέσματα σε έναν βαθμό να υλοποιήσουμε ήδη. Και για την άλλη ερώτηση κυρίας, η παρατήρηση κυρίας Γελαζάντερ ότι δεν είναι πάντα οι καλοί αυτοί που φαίνονται καλοί, ότι μέσα αυτούς κρύβονται και κάποιοι κακοί ή μέσα στους κακούς είναι και κάποιοι που στην πραγματικότητα είναι καλοί. Δηλαδή ότι τα αποτελέσματα εν τέλει και όταν μπορούμε να, δώσουμε, να κάνουμε μια ανασκόπηση με βάθος χρονικό στο παρελθόν 7-8 ετών, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά από αυτό που περιμέναμε. Και έστω, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καθαρή ανάλυση και όποια ε, δήλωση εκδίδουμε να είναι για μας αξιόπιστη για να διαφυλάξουμε και το κύρος του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν θα επιτρέψουμε να μας παρασύρει ο σε δηλώσεις οι οποίες είναι αμφιβόλου ποιότητας ε, ή εν πάση περιπτώσει αμφισβητήσιμες. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό το αποκλείω για οποιοδήποτε συνάδελφο από το ελεγκτικό συνάδελφο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο είμαστε πάλι εδώ σε, σε μια δεύτερη έκθεση για το 2018 ως προτεραιότητα ναι αλλά όχι ως ύψιστη προτεραιότητα παρακολουθούμε το θέμα περαιτέρω. μας ενδιαφέρει για τον κύριο Σαλαφράνκα που αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και την έμφαση που δίνεται στα, σε νέα θέματα. Ναι, το γνωρίζουμε και σε προηγούμενα έτη και φέτος μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα ότι δηλαδή ε, υπάρχουν πλέον νέα καθήκοντα τα οποία δεν ε, βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν άμυνα και ασφάλεια παραδείγματι, καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραδείγματι ή μετανάστευση. Είναι ζητήματα που στο παρελθόν δεν είχαν παρουσία, δεν, ε, δεν έπαιζαν κάποιο ο ρόλο στην ε, πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η διαδικτυακή ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα και σε κάθε κατάσταση βεβαίω μπορεί οι εξελίξει να μα ε, καταλαμβάνουν εξαπίνηση, να μην είμαστε πάντα σε θέση να προβλέπουμε εξελίξει και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να προετοιμαστούμε καλύτερα για να καλύπτουμε νέου τομεί δραστηριοτήτων. Αναφέρεστε σε αλλαγέ δεδομένων ε, και αρμοδιοτήτων ε, ότι πλέον δηλαδή δεν είμαστε στον παραδοσιακό σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε την πολιτική γειτονία, έχουμε το θέμα της μετανάστευσης που όλο και μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζει. Έχουμε όλο και περισσότερους ε, συναδέλφους του Ελεκτικού Συνέδριο που εξειδικεύονται στα θέματα αυτά και βεβαίως πάντοτε προσπαθούμε και το προσωπικό μας να το προσαρμόζουμε, προσαρμόζουμε τις αξιότητες τους, τις νέες αρμοδιότητες και βεβαίως και ποιοτικά είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι. 47 ήταν οι συστάσεις μας ε, για το πρόγραμμα εργασίας του 2018, αυτές που έχουμε προβλέψει, 50 να το στρογγυλέψουμε. με διαφορετικό βέβαια format κάθε φορά, αλλά αυτό έχει να κάνει με το πρόγραμμα και το επίπεδο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε, δηλαδή του προηγούμενου έτους και πάλι. Η στόχευσή μας είναι να περνούμε, όχι τόσο, να, περνούμε περισσότερο από την συμμόρφωση στις επιδόσεις, από το compliance στο performance, γιατί αυτό νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία και έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη ένταση εργασία. Και όσο καλύτερη είναι η συμμόρφωση των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο περισσότερο μπορούμε εμεί να στραφούμε στι εκθέσει μα, ε, στι επιδόσει, στο performance κατά τα άλλα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως προς τους ανθρώπινους πόρους όπως και κάθε άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώμεθα από τις πολιτικές αποφάσεις αυτή τη στιγμή πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ισχύουσα απόφαση για περιοικοπές τη δαπάνε προσωπικού κατά 5% που ισχύουν για όλους προφανώς και εμείς το τηρούμε. Καταβάλουμε προσπάθεια για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε καλό δρόμο. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι αυτά ε, τα νέα και φιλόδοξα καθήκοντα που αναλαμβάνουμε πρέπει να εκτελεστούν με το υφιστάμενο προσωπικό. Αυτό σημαίνει αναδιαρθρώσεις για να, ζητήσουμε, για να επιτύχουμε το στόχο της αποτελεσματικότητας και βέβαια εν και του Brexit δεν φαίνεται να βελτιώνει την κατάσταση, μάλλον θα επιδεινωθούν οι δυσκολίες. Πάντως εμείς πάντοτε προσπαθούμε να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα ώστε να ερώμεθα στο ύψος των απαιτήσεων. Η κυρία Λαβάκοβα μίλησε για τις σχέσεις μεταξύ των κοινοβουλίων. Εγώ εκπροσωπώ το Ελεκτικό Συνέδριο εδώ και πέντε χρόνια από την αρχή ήδη ε, της ανάληψης των καθηκόντων μου, 12-13, ξέρετε πριν ήμουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, παρακολουθώ τις σχέσεις αυτές, ε, βελτιώνονται διαρκώς, μπορώ να το επισημάνω αυτό. Και βεβαίως το ορίζει και ο κανονισμός ότι κύριος εταίρος μας, συνομιλητής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, αυτό που ονομάζω Πόρτο Βέντρι. Είναι το πρώτο σημείο επαφής, επικοινωνίας, είναι εκεί που στενόμαστε σαν στο σπίτι μας. Είναι ε, ο τόπος διαμονής και κατοικίας του Ελεκτικού Συνοδρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά βέβαια στο performance reporting πρέπει οπωσδήποτε και να δούμε και τη συνέπεια σχέση με τη διοικητική εφαρμογή, αλλά και τη βελτίωση της νομοθεσίας για το μέλλον. Και η βελτίωση της νομοθεσίας για το μέλλον ε, είναι αρμοδιότητα των επιμέρους των λεγόμενων τεχνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και εδώ σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το τμήμα των εκθέσεων που έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις θα έχουμε επικοινωνία όχι μόνο με εσάς αλλά και με τις επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ε, έχει ιδιαίτερα κάνει προσπάθεια και το ελεκτικό συνέδριο για βελτίωση των επαφών και βέβαια με την διάσκεψη των Προέδρων που έχει βοηθήσει ιδιαίτερα και νομίζω ότι στο μείζον τμήμα των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουμε πολύ καλές επαφές. Όχι με όλες, δεν θέλω κανέναν να κατηγορήσω ή να αναφέρω κάποιο όνομα, αλλά βλέπουμε και όποιος έρχεται στις επιτροπές σας γνωρίζει ότι υπάρχει για ορισμένες αρμόδιες για νομοθετική δραστηριότητα, για νομοθέτης ε, επιτροπές, κάπου, κάπου υπάρχουν ελλείμματα. Έχουμε εδώ τον συνάδελφο μαζί στην ομάδα μας, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις επαφές με την κοινοβουλευτική πλευρά. Εμείς λοιπόν κάνουμε κινήσεις, αλλά πρέπει και από την άλλη πλευρά η αποδοχή να βελτιωθεί και χωρίς να μου αρέσει καθόλου η διατύπωση, μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι χρειάζεται να, κάνουμε, να, ε, χρειάζεται να γίνει ένα εσωτερικό lobbying, να, στηθούν, να σκηθούν εσωτερικές πιέσεις για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση από πλευράς του Κοινοβουλίου. Από το 12 όπου ανέλαβα εγώ και με τον προκατοχό μου. Είχαμε την πρώτη πρόσκληση της Προέδρου της Δεσκέψεως ε, των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και ε, τώρα πλέον την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηνα εγώ τη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Νομίζω ότι δείχνει μια εξέλιξη διαρκή και θετική. Θέλω να την τονίσω και ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για τη βοήθεια. Ο κύριος Σαρβάμα... είπε ότι λυπάται που δεν ήταν στην αρχή της ε, παρέμβασής μου εδώ. Ναι, ξέρω πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα. Είναι σαν το χόκεϊ επιπάγου. Έρχεται ο επιθετικός, μία, δύο, τρεις, μετά πρέπει να βγει, μετά ξαναγυρνάει. Εντάξει, ξέρουμε πώς δουλεύουν ε, οι επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Ε, τώρα για τα σημεία έμφασης είναι αρκετά, τα, είναι ορατά πιστεύω ιδιαίτερα το θέμα της γεωργίας, ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα της μετανάστευσης έχει ιδιαίτερη σημασία όπως και της ασφάλειας, ε, ε συναφές. γενικά ό,τι έχει να κάνει με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, περιφερειακή πολιτική επί δηλαδή θέματα τα οποία θα έχουν σημαντικό ρόλο και στη διαπραγμάτευση του πολίτου δημοσιονομικού πλησίου. Αντίστοιχα, ενδιαφέρουν και εμάς και θα αντικατοπτριστούν και στο πρόγραμμα εργασιών μας. Μιλάτε για συγκεκριμένη αξιολόγηση, μιλάτε για βελτίωση των εκθέσεών μας. Νομίζω ότι εδώ και καιρό έχει αρχίσει η επισκόπηση των συστάσεων και τη υλοποίηση των συστάσεών μας και προκειμένου να ε, βελτιώσουμε την ε, διατύπωση και τη δική μας συνεισφορά να κάνουμε αυτό που λέμε fine tuning. Δηλαδή κοιτάμε να δούμε από τις συστάσεις μας τι μπόρεσε να περάσει, τι είναι κατανοητό και τι χρειάζεται εμείς να βελτιώσουμε. Και εδώ πιστεύω ότι πρέπει πιο συγκεκριμένα να παρακολουθούμε την ε, εκτέλεση, την προσαρμογή στις δικές μας συστάσεις και να βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και διατυπώνουμε τις δικές μας συστάσεις και ε, αναλύσεις. Αυτά για να γίνονται βέβαια και καλύτερα κατανοητές. Νομίζω ότι έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. And I thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους. Ίσως ε, υπάρχουν κάποιες προσθέσεις ερωτήσεις από την κυρία Γιάλα Ναι, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Λένε ότι συμφωνώ ότι έχει βελτιωθεί η σχέση με τα υπερκετακατά κατά που είχαμε. Θα ήθελα όμως να σας εκφράσω και μια βηθιά ανησυχία που έχω σε σχέση με την ε, οικοδόμηση του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι να χρησιμοποιηθεί το λεκτικό συνέδριο και εκθέσεις του να, ως βάση για να αιτιολογηθούν περικοπές. Όπως είπε και ο κύριος Σελαφράνκα, το έργο του ελεκτικού συνεδρίου και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον αριθμό των επιτροπών που σας έχουν προτείνει διάφορα θέματα ή έχουν ενδιαφέρον ε, να τους βοηθήσετε. Όμως, απ' την άλλη ανησυχώ, μήπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως εργαλείο Και επειδή κανένας δεν θέλει να είναι ο κακός ε, τέλο πάντων στην ταινία, μπορεί να ε, χρησιμοποιήσει τις εκθέσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου για να νικήσει τον εχθρό. Μας μένει 1,5 χρόνος ε, στη θητεία. Εσείς είπατε ότι είσαστε πολύ προσεκτικός έτσι ώστε να μας βοηθήσετε στο να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. και θα ήθελα να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτήν την μάχη. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εκθέσεις ως εργαλείο, γιατί δεν θα βοηθήσει καθόλου ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Ελεκτικό Συνέδριο κάτι τέτοιο. Ε, εσείς ε, αναφερθήκατε σε μια μερική ε, ανανέωση. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε το μέλλον αυτής της ανανέωσης, δηλαδή σε σχέση με την ε, κατάσταση στο ελεκτικό συνέδριο και αν μπορούμε να περιμένουμε η βελγική κυβέρνηση να λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου ή όχι. Παρακαλώ να απαντήσετε συντομία. Όταν θέλουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, αυτό δεν ε, το κάνουμε μόνο για τον, ε, λέγοντας ότι ο προπολογισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Η δική μας προσπάθεια είναι ο όσα ε, κονδύλια προβλέπονται στον προπολογισμό να χρησιμοποιηθούν σκόπιμα, χρηστά. Αν κάποιος δηλαδή έρθει και πει ότι αυτά τα κονδύλια είναι άσκοπα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να δοθούν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, τότε σίγουρα δεν θα το πει με την νομοποίηση του ελληνικού συνεδρίου, γιατί αυτό είναι και το νόημα του όλου δημοσιονομικού πλαισίου, το εύρος των δαπανών των, ε, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζεται για 7 χρόνια. Και εμείς ε, ε, δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λόγο να κόψουμε αυτά, να μειώσουμε αυτά τα κονδύλια. Το θέμα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε χρηστά για να μπορούμε να έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν πολιτική απόφαση το πόσο υψηλά θα είναι αυτά τα ε, κονδύλια. Δεν είναι απόφαση του ελεγκτικού συναδρίου. Το αποφασίζει το Συμβούλιο Υπουργών από κοινού το Κοινοβούλιο σε μια διαδικασία συναπόφαση. Δεν έχουμε εμεί κανένα ρόλο να παίξουμε σε αυτή την απόφαση. Εμεί το μόνο που έχουμε να φροντίσουμε είναι αν αυτά τα κονδύλια όντω είναι σκόπιμα και έχουν δαπανηθεί ε, όπω πρέπει. Βεβαίω πάντα μπορεί κανείς να πει ότι ε, υπήρξαν ε, ε, ε, καταχρήσεις, αλλά το θέμα είναι και εμείς πώς διατυπώνουμε τις απαντήσεις μας σε αυτές τις κατηγορίες. Σε σχέση με αυτό που είπατε για τις έρευνες που βρίσκονται να εξελίξει δεν μπορώ να σας πω κάτι. 100% όμως μπορώ να σας πω ότι γίνεται δυνάμει των κανόνων που έχουν συμφωνηθεί. Η περίπτωση λοιπόν των πληροφοριοδοτών διεξάγεται κανονικά, τα δεδομένα έχουν πάει στην ε, Όλαφ. Η Όλαφ ε, έκανε τις ε, έρευνές της, συνεχίζει να ερευνά. Υπάρχει βεβαίως η αρχή της αθότητας καταρχήν και εξετάζονται τα στοιχεία. Υπάρχουν δύο δυνατότητες, τα είπα και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια ε, συνέντευξη τύπου. Είτε θα κλείσει η υπόθεση, είναι μια επιλογή, η άλλη είναι ότι θα υπάρξουν ε, ποινές. Είναι σαφές το πράγμα. Αυτά μπορώ να σας πω σήμερα ως προς αυτό. Παραπάνω δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Και όλα, ξαναλέω, γίνονται ε, κανονικά με τους, ε, σύμφωνα με τους ε, κανόνες. Και βεβαίως τηρούνται πλήρως και οι διατάξεις που αφορούν στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών. Αν, υπήρχε κάποια διαρροή, βεβαίως θα υπήρχαν σοβαρές απειλές, σοβαρές συγγνώμη. Πάντα έχουμε κανόνες τους οποίους φροντίζουμε να τηρούμε. Αυτά ως προς αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο στη στιγμή αυτή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για το πρώτο ερώτημα της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, Εμεί ω ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα είμαστε καλοί θεματοφύλακε για να, υπάρχουν, ε, για να υπάρχουν μάλλον καλές σχέσεις ε, έτσι ώστε με τι επιτροπέ τη τεχνική του Κοινοβουλίου για να μπορούμε να σα βοηθήσουμε και εσά να κάνετε τη δουλειά σα. Ευχαριστώ. όλου. ευχαριστώ εσά και του συναδέλφου σας από το Ελεγκτικό Συνέδριο που ήσασταν σήμερα εδώ. Κλείνουμε λοιπόν την δημόσια συνεδρίαση και θα σα δούμε αύριο το πρωί στι 9. Καλό σας βράδυ.